Θα ήθελα να αρχίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι ε, με το σημείο 4 όπως αποφασίσαμε χθε, ε, που είναι η γνωμοδότηση της Ελίζαπετ Σρέτερ για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να δώσω λόγο στην Ελίζαπετ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφε με ήττα μάλλον, διότι δεν βλέπω και πολλούς συναδέλφους γύρω-γύρω. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι η ιδέα της έκθεσής μου, της γνωμοδότησης καλύτερα. Είναι ένα στοιχείο του πακέτου που συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε χθες. Γιατί για πρώτη φορά τώρα, σε αυτό τον τρόπο και με αυτή τη μορφή, Έχουμε μια κοινή ομπρέλα, μια κοινή στέγη για τα ταμεία που ξαναμπήκε η ανάπτυξη της υπαίθρου. Το είχαμε στο παρελθόν σε μερικές περιφέρειες, στις ιδιαίτερα μειονεκτικές, μετά εγκαταλείφθηκε και τώρα ξαναμπήκε σε αυτή την κοινή ε, ρύθμιση. Αυτό το θεωρώ θετική εξέλιξη. Και γι' αυτό εξίσου είναι σαφές ότι θα πρέπει να κοιτάξει η συγκεκριμένη έκθεση αυτό το σημαντικό στοιχείο ε, της περιφερειακής πολιτικής και της ανάπτυξης υπαίθρου να ε, είναι καλά προσαρμοσμένο αυτό το στοιχείο εκεί που έχει ενταχθεί, δηλαδή να ε, ταιριάζει σωστά. Αυτό είναι από τα σημαντικότερα της έκθεσης. Είναι νομοθετικού περιεχομένου, αλλάζουμε δηλαδή το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάνουμε και κάποιες μικροδιορθώσεις. Γενικά συμφωνώ με το πνεύμα του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει σωστή κατεύθυνση και αναπτύσσει ε, και μεταξελίσσει μάλιστα τον ισχύοντα ε, κανονισμό και έχει την πρόθεση ε, μαζί με τα άλλα ταμεία να επικεντρώσει τις δραστηριότητες στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. και βεβαίως και τις μεταρρυθμίσεις κοινή γεωργικής πολιτικής. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο κεντρικά πακέτα και της ανάπτυξης πέθρων, Δηλαδή είναι και στα δύο αυτό, δεν είναι μόνο στη γεωργία. Από τη μια θα πρέπει έχουμε τη γενική ανάπτυξη, αλλά δεν θα πρέπει η κοινή γεωργική πολιτική και η ανάπτυξη της υπαίθρου ε, να αλληλοανερούνται. Δηλαδή, τι εννοώ, έχουμε έξι ε, βασικά σημεία σε αυτό το μέσον και αν τα μελετήσει κανείς από τα έξι αυτά τα τέσσερα είναι ε, πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα με την κοινή γεωργική πολιτική. Ένα άλλο είναι μισό-μισό, δηλαδή ε, μισό έχει ε, ε, μεγάλη περιφερειακή επίπτωση και το άλλο μισό έχει να κάνει με την παραγωγή ενός αγροκτήματος. Και για την ανάπτυξη της υπαίθρου, το τελευταίο, το έκτο, είναι αποκλειστικό ε, θέμα ανάπτυξης τη υπαίθρου και δεν συνδέεται με τη γεωργική παραγωγή σε ένα αγρόκτημα ή σε μια εκμετάλλευση. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα μέσο της περιφερειακής πολιτικής και το εντάσσουμε πλήρως εκεί. Έχει και σχέση και με τη γεωργία. Γιατί το αναλύω τόσο πολύ, διότι υπάρχει ένα ζήτημα τώρα κομβικό σε τούτη εδώ την Επιτροπή, την Περιφερειακή, που συνδέεται άμεσα. Και αυτό είναι το Το είδαμε και χτες ε, στην ψηφοφορία. Θελήσαμε ρητά να υπάρχουν τρεις κατηγορίες περιφερειών. Οι μειονεκτικές περιφέρειες, οι μεταβατικές περιφέρειες και οι πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αυτό δεν φαίνεται τόσο πολύ στο μέσο ανάπτυξη της υπαίθρου και ακούστηκαν πάρα πολλές ε, παρακλήσεις και αιτήματα να υιοθετηθεί και εκεί. Μπορώ να το καταλάβω απολύτως. Εάν δούμε τι λέει η πρακτική και έχει να κάνει και με τη συγχρηματοδότηση και τα ποσοστά της είναι πάρα πολύ ε, ε, δύσκολο να έχεις διαφορετικά ε, συστήματα και διαφορούς συντελεστές για τη συνυπευθυνότητα και τη συγχρηματοδότηση. Είναι πάρα πολύ αλληλένδετα όλα αυτά. Και έχουμε δυσκολία, διότι στη Γεωργία οι συντελεστές συγχρηματοδότησης δεν προσανατολίζονται στις περιφέρειες, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχθεί το γεωργικό εισόδημα. Και εκεί έχουμε τεράστια σύγκρουση και μάλιστα ένα άλλο το πρόβλημα. Εγώ βρήκα μια λύση ε, που πιστεύω ότι μπορούν όλοι να μείνουν ικανοποιημένοι. Διότι έχουμε και δύο άλλες απαιτήσεις. Ε, θέλουμε τους ίδιους συντελεστές ε, με τα περιφερειακά μέσα και για την ανάπτυξη της Βέθρου, γιατί αλλιώς έχουμε τεράστια σύγκρουση και δεν μπορούν να κουμπώσουν μεταξύ τους τα ε, ταμεία. Δεν μπορείς να έχεις για το κάθε μέτρο διαφορετικό συντελεστή. Και όταν έχουμε και από πολλά ταμεία χρηματοδότηση, καήκαμε. Γι' αυτό ε, έχω κάνει αυτή την πρόταση, αλλά ως εναλλακτική επιλογή. Σας είπα είναι έξι τα βασικά σημεία και ε, το ένα μόνο αφορά αμυγός αυτή την ιδιαιτερότητα και ένα άλλο ή μάλλον μισό άλλο. Ε, πώς θα τα συγκεράσουμε όλα αυτά, γιατί οι υπόλοιποι συντελεστές υπολογίζονται τελείως διαφορετικά. Ανάλογα με την γεωργική παραγωγή. Αν έχω μια εκμετάλλευση στο βουνό, ας πούμε, είναι αλλιώς η παραγωγή μου από το αν έχω στην πεδιάδα ε, τεράστιες εκτάσεις, εκτάρια. Ε, γι' αυτό βρήκα μια λύση η οποία ε, λέει το εξής. Τα κράτη-μέλη έχουν την επιλογή. Γιατί χρειάζεται αυτό, διότι ακούμε και από τις μεταβατικές περιφέρειες το αίτημα που λέει ότι δεν θέλουμε προσαρμοσμένα ποσοστά, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε λιγότερα έργα. Εμείς θέλουμε πολλά μικρά έργα και ε, χρηματοδοτικά γίνεται αυτό μόνο αν παραμένει χαμηλός ο συντελεστής. Έχω βάλει λοιπόν μια πρόταση. Τα κράτη-μέλη που θέλουν να έχουν τους ίδιους ε, συντελεστές, γιατί είναι καλύτερο για τα διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πολλά ταμεία, μπορούν να το κάνουν. Γιατί είναι περιορισμένα τα χρήματα. Ε, το δέχονται να έχουν λιγότερα έργα, δεν τους πειράζει. Αλλά εκείνοι που λέγουν ότι θέλουμε να έχουμε πολλά μικρά προγράμματα και να το κατανείμουμε αυτό το ποσό σε πολλούς δικαιούχους, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει για την περιφερειακή μας ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και θέλουμε να το συνδέσουμε με την παραγωγή στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αυτοί μπορούν να το πράξουν. Δηλαδή είναι επιλογή. Και ε, έχω προτείνει αυτή τη λύση στους συναδέλφους του ΕΛΚ. Υπάρχει δυνατότητα ε, τα κράτη να διατηρούν τους ίδιους συντελεστές φαντού, ε, αλλά και εκείνα τα κράτη που θέλουν να επιλέξουν μια άλλη λύση γιατί έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης και από τον κρατικό κόρβανα, μπορούν. Νομίζω είναι ιδιώδης λύση για να φτιάξουμε εδώ μια γέφυρα. Ένα τελευταίο. Έχει ένα κέντρο βάρους η έκθεση και η γνωμοδότηση είναι και λογικό άλλωστε αυτό, οι ομάδες leader, η μέθοδος του leader δηλαδή. Έχουμε και πιο στενή σύνδεση με το γενικό κανονισμό και από το άρθρο 28 μέχρι το άρθρο 31 του γενικού κανονισμού ε, έχουμε υιοθετήσει τη μέθοδο leader απλώς εξειδικεύεται σε αυτό τον κανονισμό και δική μου δουλειά ήταν να το προσαρμόσω ε, αναλόγως. Αυτά τα βασικότερα. Γιατί επιλέγουμε τη μέθοδο Leader, διότι προέρχεται από την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πάνω από 20 χρόνια έχει γνωρίσει απόλυτη επιτυχία, τεράστια, και γι' αυτό το βάλαμε και στο γενικό κανονισμό, διότι θεωρούμε ότι μπορεί να ισχύσει και για πρωτοβουλίες δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά και για, άλλα, και το, πώς το για τις πόλεις, για την αστική διάσταση. Τώρα όμως έχουμε και μια πολύ μικρή δυσκολία στον κανονισμό που είναι όμως ε, σοβαρή και μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Το έχω συζητήσει εκ των προτέρων και με τους κοιόδης ηγητές. Και αυτό είναι το πώς ορίζεται η ύπεθρος. Ορισμένοι δεν θέλουν καθόλου ορισμό. Εγώ το θέλω. Γιατί θέλω ανάπτυξη της ύπεθρου. Ε, και πώς ορίζεται η ύπεθρος. Δεν υπάρχει πλήρη διαχωρισμός και απόλυτο από εδώ η πόλη, από εδώ η ύπεθρος. Δηλαδή άμα πα ένα μέτρο πιο εκεί στην πόλη. Πώ θα ορίσει την ύπεθρο. Μην είναι η κάμπη. Όχι. Δηλαδή οι αγρότες που πάνε στην πόλη και πουλάνε στη λαϊκή ε, και έχουν ένα πάγκο, ο πάγκος δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ανάπτυξη πέθρου, θα πρέπει να πάνε στην πολεοδομία ή δεν ξέρω σε κάποια υπηρεσία της πόλης για να επιδιτωθούν. Ε, εδώ μιλάμε για λειτουργικούς χώρους λοιπόν, όχι αμυγός εδαφικούς. Ε, θα το βρείτε σε διάφορες τροπολογίες. Αυτά είναι τα σημεία που θεώρησα ότι ήταν τα σημαντικότερα, τα βασικά, για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το στοιχείο της ανάπτυξης υπαίθρου και να λειτουργήσει και να μην παραγωνιστεί από τις δύο άλλες μεγάλες πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης από το ΕΛΚ. Ο κύριος Σικέρσκι. W φιλάρου drugiego filaru wspólnej polityki rolnej przewidziano realizację wielu działań służących zwiększeniu Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ε, πολιτικής μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη πόρη με ταυτόχρονη ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, καταπολέμησης, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της υπαίθρου. Άρα οι στόχοι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολύ φιλόδοξοι ενώ τα μέσα που διαθέτουμε πολύ ανεπαρκή αν χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από διάφορα ταμεία θα μπορούσαν να διευκολυνθούν τα πράγματα και να προωθηθούν όλα τα προγράμματα που θέλουμε να εφαρμοστούν στην Ήπεθρο να στηριχθούν από το Κοινωνικό Ταμείο ή από το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου. Υπάρχει και ο δεύτερος πυλώνας που είναι πολύ πιο σημαντικός ποσοτικά στις νέες χώρες μέλη που πρέπει ακόμη να κερδίσουν το χαμένο χρόνο ιστορικά. Και υπάρχει και το θέμα του πρασινίσματος που πρέπει να κάνουν. Άρα η ανταγωνιστικότητα της υπαίθρου είναι χαμηλότερη εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών μελών, ούτε τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ότι το σύστημα πρέπει να είναι όσο διαφανέστερο γίνεται. Όταν κανείς υποβάλει την αίτησή του και πάρει τη χρηματοδότηση, όλα αυτά πρέπει να είναι διαφανή ώστε αυτός που ωφελείται να γνωρίζει ποια απλά βήματα πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει λοιπόν επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα είναι όλα αυτά σωστά σχεδιασμένα. Παραδείγματος χάρη καταθέσαμε την τροπολογία 10 και την, τη 40 και τη 45 για το στόχο αυτόν. Ό,τι προγράμματα μπορούν να στηριχθούν από διάφορα ταμεία, από διαφορετικά ταμεία, δεν πρέπει να απαιτούν για την εφαρμογή τους πιο πολύπλοκες αιτήσει επειδή θα χρηματοδοτούνται από διαφορετικά ταμεία. Αυτό με ανησυχεί και φοβάμαι μήπως μερικά προγράμματα τελικά δύσκολα εφαρμοστούν και καθόλου. Δεν θα υποστήριζα μια λύση που θα πρόβλεπε ένα πρόγραμμα ή ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από διαφορετικά ταμεία μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου να δυσκολεύεται στην εφαρμογή του από το γεγονός αυτό. Γι' αυτό καταθέσαμε και άλλες τροπολογίες για τη χρήση διαφορετικών ταμείων για το ίδιο πρόγραμμα ή σχέδιο. Τώρα το πρόγραμμα Leader. Υπάρχουν κανόνες και ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για τοπική διαχείριση. Υπάρχουν κανόνες για τα σχέδια leader στο άρθρο 42 ή 45 και οι κανόνες αυτοί πρέπει να ερμηνευτούν μαζί με την ισχύουσα νομοθεσία, την υπόλοιπη ισχύουσα νομοθεσία και ιδίω την τα ό,τι προβλέπεται δημοσιονομικά για την ΚΑΠ, γιατί το κύριο πρόβλημα στην εφαρμογή των προγραμμάτων Leader είναι η σύγχυση ως προς τη διαχείρισή του. Ιδίως ως προς το ποια θα είναι η διαχειριστική και ποια η πληρωτική αρχή. Αν η προσέγγιση μας είναι αυτή, τότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει και συντονισμός ως προς τα κριτήρια και τους όρους χρησιμοποίησης των διαφόρων ταμείων. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο πρέπει νομίζω να τονίσουμε περισσότερο την τοπική διάσταση. Οι τοπικές αρχές να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τοπική στρατηγική και να στηρίζουμε ακριβώς αυτούς που τοπικά εφαρμόζουν τα προγράμματα. Έχουμε και άλλες τροπολογίες, την 14, ε, την 82 και μερικές άλλες που συμπεριλαμβάνουν το 10% ορίου στήριξης που νομίζω ότι πρέπει να μεταφερθεί στο leader. Υπάρχει επίσης η πρόταση το 40% να δοθεί στο πρασίνισμα στα πλαίσια του Natura 2000 και υπάρχουν και συνδέσεις με την οδηγία για τα ύδατα. Τα μισά χρήματα δηλαδή θα διατεθούν σε μόνο δύο τομείς και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Για όλα τα υπόλοιπα, όπως την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη της υπαίθρου, θα στηρίζονται μόνο από το υπόλοιπο 50% λάθος μου φαίνεται αυτό. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά τουλάχιστον το 10% να χορηγείται. Αυτό το λέω στην τροπολογία 46 γιατί αυτό το βρίσκω περιοριστικό και νομίζω ότι πρέπει πάντοτε η κατανομή να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Επίσης αυτό το όριο του 10% στα πλαίσια του leader είναι πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό. Ήδη είναι δύσκολη η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο το 5% εφαρμόζεται, ενώ στη νέα προγραμματική 2,5%. Αυτό προτείνουμε. Και πολύ λίγες χώρες μέλη και αυτό το 5 και 2,5% θα μπορέσουν καν να το χρησιμοποιήσουν. Τώρα για τους ορισμούς και τις έννοιες. Ορισμένοι ορισμοί νομίζω είναι ασαφείς και δεν φτάνουν στην απαραίτητη λεπτομέρεια. Παραδείγματο χάρη η σύνδεση μεταξύ των αστικών περιοχών και της υπαίθρου Οι 16, 20, 21, 25 αυτές οι τροπολογίες αφορούν αυτό το θέμα. Ελπίζω να ληφθούν σοβαρά υπόψη αυτά που σας είπα και θα σας στείλω τις τροπολογίες σύντομα. Ευχαριστώ, δεν βλέπω κανένα άλλο σκιώδη. Όποιος θέλει λοιπόν να πάρει το λόγο. Ο κύριος Βλάσακ αν δεν απατώμε. Και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που άκουσα, τη σημαντική αυτή γνωμοδότηση δηλαδή για συμπλήρωση αυτών που ψηφίσαμε χθες. Θα ήθελα να σχολιάσω μερικά πράγματα. Πρώτον, τη φιλοδοξία να ορίσουμε καλύτερα τι ακριβώς είναι οι υπεθρος και οι υπαίθριες περιοχές έχουμε ορίσει σχετικά καλά τι είναι αστικές περιοχές και τελικά από την παλιά μου έκθεση είχαμε συμφωνήσει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε πανενοσιακώς τι είναι ακόμη και αστική περιοχή. Γιατί διαφέρουν οι ιστορικές και φυσικές ιδιότητες από χώρα σε χώρα. Το ίδιο ισχύει και για την Ήπεθρο. Πρέπει να το δούμε λειτουργικά Από ό,τι ξέρω και καταλαβαίνω η έννοια αυτή της λειτουργικής περιοχής πρέπει να περιέχει ένα κριτήριο ποιότητας της ζωής όσων ζουν εκεί. Μία λειτουργική περιοχή δηλαδή πρέπει να λειτουργεί σωστά. Για τη μέθοδο leader ξέρω ότι θεωρείται πολύ σωστή και χρησιμοποιείται ευρέως αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστεί και να χρηματοδοτηθεί. Γι' αυτό τη στηρίζω και εγώ, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μέχρι τώρα ήταν πολύ χαμηλότερη η χρηματοδότηση που χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο, τη μέθοδο leader. Αν αυξηθεί η χρήση της θα γίνει και πιο δύσκολη η εφαρμογή γιατί θα αυξηθεί και το, λειτουργικό, το διοικητικό μάλλον κόστος Τέλος, για τα ίδια τα σχέδια ή προγράμματα, συμφωνώ ότι πρέπει να εφαρμόζονται από τις τοπικές αρχές. Ε, Γιατί τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια πρέπει από εκεί να εφαρμόζονται για να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής που ασχολείται με την ανάπτυξη της υπαίθρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Καταρχήν ευχαριστώ εξ ονόματος της Κομισιόν την Επιτροπή Περίφ του Κοινοβουλίου Ρέγγι που γνωμοδοτεί σήμερα για την πολιτική ανάπτυξη της Υπέθρου. Η Κομισιόν θεωρεί ότι το έγγραφο αυτό, η γνωμοδότηση δηλαδή, κατανοεί πλήρως τι προβλήματα αντιμετωπίζει η Ήπεθρος και την λογική των προτάσεων της Κομισιόν ταυτόχρονα. Προτείνει πολλές τροπολογίες και θα ήθελα να σχολιάσω μερικές από αυτές. Για το Λίντερ, Συμφωνώ απόλυτα ότι το Λίντερ είναι από τα σημαντικότερα νέα εργαλεία που διαθέτουμε για την προώθηση του, της τοπικής διάστασης και της προσέγγισης bottom-up. Επίσης ε, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συμπεραίνεται ότι το Λίντερ συμβάλλει αποφασιστικά στην ε, ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών. Γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει να ενδυναμωθεί αυτή η προσέγγιση μέσω πρώτων της επέκτασής της σε όλα τα ταμεία κοινής στρατηγικής μέσω της ενδυνάμωσης αυτής της προσέγγισης bottom-up, μέσω καλύτερης εκπροσώπησης των τοπικών εταίρων και τρίτον βελτιώνοντας την ποιότητα των προγραμμάτων ε, τοπικής ανάπτυξης. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου είναι το μόνο εργαλείο ε, Ταμείο Κοινή Στρατηγικής που έχει επιβάλει ελάχιστο όριο 5% δαπάνησης για το leader. Αυτό το κάναμε, το καθορίσαμε μετά από προσεκτική ανάλυση των αναγκών των χωρών μελών και των δυνατοτήτων τους απορρόφησης. Γι' αυτό πιστεύω ότι αντί να αυξήσουμε την ελάχιστη συμβολή του Λίντερ που είναι 5%. Οι χώρες μέλη που θέλουν να το πράξουν, να το κάνουν εθελοντικά. Εκτός αυτού η Κομισιόν ήδη έδωσε κίνητρα για περισσότερη χρήση του Λίντερ μέσω της δυνατότητας αυξημένης συγχρηματοδότησης μέχρι το 80%. Ως προς τις υπάρχουσες λιντερικές δυνάμεις, η Κομισιόν συμφωνεί με, τον, με την εισηγήτρια ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία που υπάρχει και να τύχουν εκμετάλλευση σε όλες οι ευκαιρίες που δίνονται. Αλλά με κάποια στρατηγική και προσαρμογή και σε μελλοντικά προβλήματα που πρέπει να αναλυθούν από την κάθε τοπική αρχή για την στρατηγική της. Επιπροσθέτως πρέπει να υπάρχει μια εξισορροπημένη διαδικασία επιλογής που να εφαρμόζεται και στις νέες και στις παλαιότερες χώρες και αρχές. Τώρα για το κλίμα και το περιβάλλον. Ο, για αυτά τα θέματα καλό είναι που βλέπουμε ότι η Επιτροπή Περίφ ε, προσέχει ιδιαίτερα φροντίζει να δει με τι τρόπους θα αντιμετωπιστεί η κλιματολογική και περιβαλλοντολογική πρόκληση στο μέλλον. Το σχέδιο γνωμοδότησης θέλει 40% τουλάχιστον των κονδυλίων από το EFRD για κάθε χώρα να δαπανούνται για θέματα κλιματολογικά και περιβαλλοντολογικά αντί για 25% όπως προτείνει η Κομισιόν ή 30% όπως προτείνει η Κομάγκρη δηλαδή η Γεωρέπ. Δεν θέλουμε όμως να γίνουν όλα αυτά επιβαλόμενα και δεσμευτικά γιατί Υπάρχει το θέμα του στρατηγικού προγραμματισμού. Μετά το 2013 τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου θα βασίζονται πολύ περισσότερο στα αποτελέσματα μάλλον παρά στις δαπανήσεις. Οι ανάγκες δαπανήσεως 25% ή παραπάνω είναι απλώς μια ρήτρα ασφαλείας και θα καθοριστεί επακριβώς στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κομισιών και χωρών μελών και δεν θα είναι μια απόλυτη επιβολή. Αλλά βέβαια το ακριβές ποσοστό που θα εφαρμοστεί θα συζητιέται κάθε φορά. Τώρα να σχολιάσω το μίνιμουμ 10% συμβολής του EFRD για τις έξι προτεραιότητες. Πιστεύω ότι το ταμείο αυτό πρέπει να χέ να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη ανάλυση της κάθε περίπτωσης και ανάγκων της κάθε χώρας για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020. Τα κονδύλια λοιπόν πρέπει να χορηγούνται με βάση τα σχεδιαζόμενα αποτελέσματα μάλλον παρά σε επιβαλόμενες και προκαθορισμένες δαπάνες, ύψη δαπανών. Επίσης σημείωσα ότι η Επιτροπή Περίφ προτείνει πολλές αλλαγές στους στόχους και προτεραιότητες για τη μελλοντική ανάπτυξη της μελλοντική υπαίθρου. Γενικότερα η Κομισιόν θεωρεί ότι οι περισσότερες από τις προτινόμενες αλλαγές μειώνουν το εύρος της πολιτικής και διαστρεβλώνουν το στόχο της. Let me, however, ε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εταιρικέ συμφωνίες, στα προγράμματα συνεργασίας υπό το Λίντερ. Για την επιχειρηματικότητα η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες και μικρότατες επιχειρήσεις. Θέλω όμως να επιμείνω ότι και πιο μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα αποκλείονται από τις στηρίξεις ιδιαίτερα ως προς τη μεταφορά γνώσης, τεχνογνωσίας, ανάλογα με το πρόγραμμα. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της υψηλότερης, του υψηλότερου ρυθμού συγχρηματοδότησης των μεταβατικών περιοχών. Αυτό φυσικά το συζητήσαμε αλλού, αλλά πρέπει και εδώ να λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα της συζήτησης εκείνης. Κάλυψα έναν μικρό μόνο αριθμό των θεμάτων που τίθενται, αλλά ελπίζω να σας έδειξα ότι η Κομισιόν παίρνει πολύ σοβαρά τη δουλειά της Επιτροπής Περίφ ως προς την ανάπτυξη της υπαίθουρου και προσβλέπουμε σε περισσότερη και καλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Um, I would like, I don't know, Elizabeth, would you like to, to make, but very brief comments. Θα ήθελα να κάνω μερικά σύντομα η Ελίζα αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Τρία πράγματα. Πρώτον, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι αναγνωρίζει τις υφιστάμενες ομάδες leader, βεβαίως, αλλά θα πρέπει να εγκριθούν τα νέα τους έργα πριν πάρουν καινούργια χρήματα. Έτσι δεν είναι. Θα το κοιτάξω, θα το μελετήσω και θα δω μήπως χρειάζεται αλλαγή διατύπωση. Είναι γεγονός, αυτό εννοούσα. Δεν θέλω αυτόματη αναγνώριση, αλλά δεν θέλω να ξαναστηθούν αυτές οι ομάδες. Υπάρχουν ήδη. Αν υπάρχουν καλές ιδέες, καμία αντίρρηση. Θα το ξανακοιτάξω και θα προσπαθήσω να βοηθήσω να βελτιωθεί η διατύπωση. Εγώ πήρα τη διατύπωση όπως είχε. 20 χρόνια τώρα πηγαίνει καλά αυτή η δουλειά και υπέθεσα ότι και τα επόμενα χρόνια θα πάει καλά. Κατά την άποψή μου αυτό το γράφω. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το κοιτάξουμε. Το δεύτερο, γιατί αύξησα ε, το ποσοστό των πόρων, ε, των φυσικών πόρων, γιατί είναι αρμόδιο όργανο εκεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος και εγώ υιοθέτησα τη θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Για τις μεταβατικές περιφέρειες Νομίζω ε, αυτό που πρότεινα βρίσκει σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λύσαμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο και ελπίζω να γνωρίσει και την υποστήριξη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν και το σημείο 4 και θα πρότεινα να ε, ορίσουμε προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Είπαμε 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι είναι. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να περάσουμε στο επόμενο θέμα να δείξουμε λίγη ευελιξία όμως γιατί ο Μάρκος πρέπει να φύγει να πάει να ψηφίσει κάπου σε άλλη επιτροπή. Λοιπόν, ερωτώ ποιος θέλει το λόγο για το ε, μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, τη διευκόνηση αυτή. Μαζί με τους σκιώδεις για να κανονίσουμε λίγο την πορεία μας χρονικά. Δεν βλέπω το σκιώδη μας. Όλοι εσείς θέλετε να μιλήσετε και ο Μάρκος Πίπε. 11 ε, παρατέταρτο. Πρέπει να το αναβάλουμε. Δεν προλαβαίνει σε 5 λεπτά. Πρέπει να φύγει ο Μάρκος να πάει να ψηφίσει σε άλλη επιτροπή. Στην Ήτρε, αν θέλετε να ξέρετε. Λοιπόν, 11 ε, παρατέταρτο. Θα συζητηθεί το θέμα το αργότερα, σε μία ώρα. Το πρόβλημα όμω είναι ότι η κυρία Κλέβα είναι εδώ. Τι θα κάνουμε τώρα. Ε, so, Marcus, we have Μάρκους, έχουμε 7 λεπτά. Θες να κάνεις την παρουσίασή σου. Λείπει και η κυρία Κλέβα. Τι να κάνω, διάλειμμα. Δεν πειράζει, αλλά δεν έχει και νόημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πάρα πολύ σύντομα. Δυστυχώ πρέπει να φύγω να πάω στην Επιτροπή Βιομηχανίας για να ψηφίσουμε ε, την ε, έκθεση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εμείς και ό,τι συγητή ζητώ συγγνώμη, πρέπει οπωσδήποτε να πάω. Εχθές ψηφίσαμε ε, τον κανονισμό για τα διορθωτικά ταμεία για το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης Το άρθρο 48 το συμβιβασμό 50 και καταργήσαμε κάποια ε, μέσα που έχουν να κάνουν με τη διευκόλυνση για την Ευρώπη, συνδέοντα την Ευρώπη. Ε, δεν ξέρω, μα έφυγε αυτό λάθο, ήτανε. Γιατί έχουμε πάρει άλλε αποφάσει σε ομάδε εργασία ε, εγκάρσει ε, και με την Επιτροπή Μεταφορών και με τη δική μα εδώ την Επιτροπή και αυτά που ψηφίσαμε τα καταργούν. Θέλω να σας θυμίσω τα σημαντικότερα σημεία, πέντε είναι. Είμαστε πάρα πολύ υπέρ αυτού του μέσου τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη ω Περιφερειακή Επιτροπή, γιατί συνδέονται πολύ σημαντικέ περιφέρειε. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση. Θα πάρουν χρήματα, αλλά εκτός του 2,5% του ΑΕΠ ε, γιατί δεν είναι δίκαιο ε, να έχεις ένα μέσο το οποίο να διαχειρίζεται κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να τιμωρούνται αν υπερβαίνουν το 2,5% του ΕΠ. Δεύτερο, προτείνω ε, ιδιαίτερη εστίαση στη διασυνοριακή συνεργασία, δηλαδή στην πραγματική μεθόριο. Κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το ρυθμίσουμε και να προτιμήσουμε τις παραμεθόριες περιοχές. Και ένα τελευταίο. Σε περίπτωση που στα πλαίσια αυτού του μέσου ε, περισσεύουν χρήματα, προτείνω ε, ένα είδος ταμείου ανακύκλωσης αυτών των ε, χρημάτων για να δαπανώνται εκεί σε αυτές τις χώρες όταν κάποιες χώρες έχουν ταμιακές δυσκολίες. Σε περίπτωση που οι χώρες το επιθυμούν βεβαίως. Αυτό το βρίσκεται και στο νομοθετικό κείμενο. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να τα αφήσω εδώ αυτό τώρα να σταματήσω να ε, φύγω και ελπίζω σε μία ώρα 11 παρατέταρτο να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να μην συζητήσουμε, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα της Πρόεδρου, το ότι μέλη γενέστε διαδικαστικά. Ελπίζω να έχετε ακόμα πέντε λεπτά. Αν φύγετε, τότε θα αναστείλουμε τη συζήτηση. Έχεις πέντε λεπτά. Ωραία, να ακούσουμε κάποιον ομιλητή. Νομίζω ότι ο Βλάσεκ είναι ένας από τους σκιώδεις που είναι εδώ. Και ο Μπαστινάρο θα έρθει και τότε θα είναι 11 παρατέταρτο. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια περίπλοκη, μήπω είναι περίπλοκη η συζήτηση. Καλύτερα θα ήταν με όλου του συναδέλφου. Εντάξει, τότε να στέλνουμε τη συζήτηση, την ε, ε καθυστερούμε μέχρι τις 11 παρατέταρτο. Από ό,τι κατάλαβα, ο Γευγένη αντικαθιστά τον Βόιτσικ Κλέβερ και είναι το σχέδιο γνωμοδότησης για τα δημοσιονομικά μέσα για τις ΜΜΕ. Έχεις το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος... Η συνάδελφος Κλέβα μου ζήτησε να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματός της γιατί δεν είναι σε θέση να σας παρουσιάσει αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης λόγω σοβαρών πολιτικών δεσμεύσεων στη χώρα της στη Σλοβενία. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέσα μέσα στο πλαίσιο του επόμενου προ... πολιτού σχεδίου ε, προϋπολογισμού. Ε, τώρα η κυρία Κλέβα έχει σχεδιάσει μια γνωμοδότηση ιδιαίτερα όσον αφορά την χρηματοδότηση των ΜΜΕ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, τον περασμένο Απρίλιο. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι, του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν ότι η αποτελεσματικότητα των δαπανών από το ΕΤΠΑ έχει παρεμποδιστεί λόγω του ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν ήταν κατάλληλο για τα διάφορα είδη μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Στο σχέδιο χνομοδότησης η συγγήτρια λοιπόν αναφέρεται σε αυτά τα πορίσματα και μεταξύ άλλων αναγνωρίζει πως αυτή η κατάσταση έχει εντοπιστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κεφάλαιο 4 για τα χρηματοπιστωτικά μέσα όσον αφορά τις ε, διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τέτοιες ε, πλατφόρμες. Επίσης θυμίζει και ζητά σαφήνεια και διαφάνεια για το νομικό πλαίσιο για αυτά τα <coughs> χρηματοπιστωτικά μέσα. Η συγκήτρια διαπιστώνει πως ε, στο νομοθετική πρόταση για την επόμενη προγραμματική περίοδο μια τέτοια έκθεση θα καταστεί υποχρεωτική υπό τη μορφή της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Όσον αφορά την έκθεση για τη αξιόπιστα συστήματα παρακολούθησης που θα είναι ειδικά για τα δημοσιονομικά μέσα, η κυρία Κλέβα είναι της άποψης ότι ενώ το δικαστήριο πιέζει για να επιβληθούν απαιτήσεις και όροι, θεωρεί πως τα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής είναι ε, προγράμματα που αφορούν τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό αυτές ε, οι διατάξεις ε, δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στην βραχυπρόθεσμη ε, κερδοφορία αλλά και στα υψηλά κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Η κυρία Κλέβα επίσης σημειώνει πως αυτή μια τέτοια έκθεση θα ήταν πολύτιμη στο τέλος της νομοθετικής περίοδου 2007-2013 και προσβλέπει στη συνεργασία με τους Κιώδης γι' αυτό το φάκελο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ να μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Για την ώρα έχω μόνο τον Λάμπερ Βανίστερο στον κατάλογο ομιλητών. Ε, αποφασίστε λοιπόν εάν θέλετε να πάρετε το λόγο. Πόσα λεπτά, όσο θέλεις. Ναι, καμιά ωρίτσα. Αφού δεν έχει εξαντληθεί από τη χθεσινή ψηφοφορία, σου επιτρέπουμε να μιλήσει μέχρι τι 10.30 άμα θέλει. Εντάξει, εγώ θα κρατήσω το χρόνο μου για αργότερα. Εγώ νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσουμε μια νέα περίοδο με νέους κανόνες αυτά τα θέματα να έχουν αποσαφινιστεί και είμαι πραγματικά ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο νέος χρηματοπιστωτικός κανονισμός, δημοσιονομικός κανονισμός με εξετάζει όλα αυτά τα μέσα και δεχόμαστε, δέχεται ότι αυτά τα μέσα που δημιουργούν τη δυνατότητα να εγγυηθούμε, να έχουμε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν χρήματα σε αυτές τις φάσεις όπου οι τράπεζες δεν παρεμβαίνουν, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν είναι νομίζω επιχειρηματικότητα, αλλά αν πας σε μια τράπεζα και αυτή σου πει όχι, γιατί κέρδη θα έχεις σε κανένα δύο χρόνια και χωρίς να είμαστε και βέβαιοι και άρα σου λένε όχι για τα λεφτά. Σε αυτή τη φάση όπου έχουμε μεγάλα προβλήματα οικονομικά πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Αλλά εδώ έχουμε την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού που δεν είναι τόσο δημιουργική τον τελευταίο καιρό, περισσότερο περιοριστική είναι. Γι' αυτό καλό είναι να βρούμε μια ανισορροπία που να μεταφράζεται μέσω του, του... κανονισμού του δημοσιονομικού και να μην συνεχίζεται αυτή η συζήτηση ε, ε, επάπειρων, αλλά να μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτά τα μέσα. Και να είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε προς την κατεύθυνση αυτών των νέων δημοσιονομικών μέσων. και να υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί. Γιατί σε κάθε χώρα, όπως ας πούμε στα προγράμματα του ΕΤΠΑ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα νέα μέσα. Όμως τα κράτη μπορούν να πούν χρησιμοποιούμε το Τζέσικα ή το ΤΑΔΕ, το ΔΙΝΑ πρόγραμμα ή τα νέα χρήματα του ΕΤΠΑ για να τα φέρουμε μέσα σε αυτό το νέο χρηματοπιστωτικό μέσο. Και ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες, ενώ άλλες όχι. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτά τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις χώρες, αλλά που δεν είναι υποχρεωτικό, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να τα χρησιμοποιήσουν. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Να μπει στις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, ώστε να πούμε εντάξει, χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες. Το άλλο ωραίο είναι ότι το εφέ μόχλευσης με αυτά τα νέα δημοσιονομικά μέσα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι επιδότησης. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει τονίσει σε διάφορα ψηφίσματα τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν υπάρχει κανείς δισταγμός από πλευράς μας. Απλά είναι το θέμα ότι πρέπει το... να έχουμε τέτοια ποιότητα διαχείρισης στις περιφέρειες και στα κράτη, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά. Mm. Πολύ συχνά δε πρόκειται για μια, ένα συνδυασμό μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην, σε κάποια περιφέρεια που συνεργάζονται με τις μικρές. Και δεν είναι απλά θέμα μικρής ή μεσαίας επιχείρησης. Και εξάλλου προς αυτή την κατεύθυνση ψηφίσαμε και χθες να μην αποκλείσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί έτσι χρησιμοποιείται όλη η αλυσίδα της καινοτομίας και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολύ συχνά στηρίζονται από μεγαλύτερες μονάδες, μεγαλύτερους ομίλους εταιριών και ή ε, πανεπιστήμια. Τονίζω λοιπόν τη σημασία αυτών των μέσων τους στόχους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα μελλοντικά προγράμματα και τονίζω και το αποτέλεσμα. Και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να επαναρχόμαστε στην Επιτροπή Προπολογισμού με ένα σωρό προβλήματα. Ελέγχου προπολογισμού με, το, με ένα σωρό προβλήματα. Ας το κάνουμε λοιπόν. Lambert, you have exhausted your speaking time for the next ε, νομίζω πως εξάντλησες ε, το χρόνο σου και το θέμα σε λίγα λεπτά. Άλλος, ο κύριος Νίλσον. Σας ευχαριστώ. Επειδή ο κύριος Βανίστερ Ρόι δεν χρησιμοποίησε όλο του το χρόνο, να πάρω και εγώ μερικά λεπτάκια. Καταρχήν πιστεύω ότι αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη με τα μέσα είναι πολύ σημαντικό καθώς και το τι δεν κάνουν. Από τη δική μου εμπειρία, στη δική μου περιφέρεια, σχεδόν πριν από 10 χρόνια προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε έναν ε, ε, περιστρεφόμενο ταμείο και προσπαθήσαμε και αγωνιστήκαμε με την κυβέρνηση για να δούμε τι ήταν νόμιμο. και τα καταφέραμε τελικά λειτουργεί και όλοι είναι ευχαριστημένοι και είδαν ποια ήταν η χρησιμότητά του. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το εκμεταλλευτούμε σε μια φάση όπου καταρα... ψιλοκαταραίει το τραπεζικό σύστημα ε, να δούμε νέα συστήματα δηλαδή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να δούμε αν ο κόσμος, ας πούμε, στη δική μου περιφέρεια ο τουριστικός κλάδος είναι πολύ μεγάλος ε, και αν θέλουμε να βάλουμε κάποια χρήματα εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα εμπειρία που είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, νομίζω ότι η Ρέιτσελ που είναι επικεφαλής ε, της μονάδας ε, χρηματοπιστωτικών μέσων ε, θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε να πάρω το λόγο εξ ονόματος της Κομισιόν. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έκανε εξαιρετική δουλειά κατά τη γνώμη μας για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Καταρχήν όπως αναφέρθηκε από τον πρώτο μιλητή συμφωνούμε πως οι νομοθετικές μας προτάσεις έχουν ε, προσπαθήσει να ανταποκριθούν στις επικρίσεις του, 10, του, συγγνώμη, του ελεκτικού συνεδρίου και ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη ενό διαφανού νομικού πλαισίου εξ αρχή για τα δημοσιονομικά μέσα. Εξάντα εξολόγηση, καλύτερε ε, εκθέσει και αναφορέ και πρέπει να έρθουμε σε επαφή ε, διαρκεί με τους συνομοθέτες για αυτό το νομοθετικό πακέτο. Επίσης, λάβαμε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης και ιδιαίτερα το θέμα της ε, μόχλευσης. Επίσης, συμφωνούμε ότι ο ορισμός ε, του, της μόχλευσης μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να λάβει υπόψη στους συγκεκριμένους στόχους, τους δικαιούχους και φυσικά την προσέγγιση της κοινή διαχείρισης. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε πως στην πράξη μπορεί να μην είναι δυνατή η μόχλευση, μπορεί να είναι αλλά ε, μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Το ε, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των ε, κοινοτικών κονδυλίων δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την κρατική, μάλλον τη δημόσια χρηματοδότηση. Θα πρέπει να παίρνει υπόψη μόνο το τμήμα του ΕΤΠΑ. 2016 δεν θα είχαμε ως, ως σημείο αξιολόγησης για να αποφασίσουμε το τελικό αντίκτυπο αυτών των μέσων. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω πώς θα περάσουμε τα σχόλια της Επιτροπής στην Μόιτσα. Ε, μήπως έχετε κάποια γραπτά σχόλια ώστε να μπορέσουμε να τα στείλουμε και να γνωρίζει και εκείνη την άποψή σας για τη γνωμοδότησή της. Ε, το μόνο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε την ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών που είναι η 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Και έτσι νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και να περάσουμε στο σημείο 18 που είναι η έκθεση, ε, η γνωμοδότηση μάλλον του κυρίου Κόβατσεφ για την ενδιάμεση έκθεση ε, για τον προϋπολογισμό για το πολιτεύσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι μια γνωμοδότηση για την ενδιάμεση έκθεση σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί θα γίνει και μια πραγματική έκθεση αργότερα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκατάθεσης, ναι ή όχι δηλαδή. Ορισμένες κυβερνήσει ζητούν την αύξηση της πρότασης της Κομισιόν για το ΠΔΠ. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να αποτύχει η στρατηγική 2020 όπως συνέβη και με τη ε, στρατηγική της Λισαβόνα το 2010. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν βασίζεται στην, ε, στην ε, νοοτροπία της κρίσης μόνο. Θα πρέπει να μειώσουμε, ότι δηλαδή πρέπει να μειώσουμε τον κοινό προπολογισμό επειδή διανύουμε μια κρίση. Το αντίθετο θα πρέπει να κάνουμε. Επίσης έχουμε θέσει τους στόχους μας μέσα στην ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020. Τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Χρειάζεται να έχουμε ψηλά στάνταρ για να εξασφαλίσουμε τους πολίτες μας. Θα πρέπει να είναι κοινή προτεραιότητα οι επενδύσεις υψηλού επίπεδου, ώστε να, να, να υπάρξει ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να παραμείνει ο βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή η πολιτική ωφελεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άμεσοι παραλήπτες καταρχήν για την ανάπτυξη και τη συμμετοχή στην ε, ενιαία αγορά αλλά και οι καθαροί συνεισφορείς στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις έτσι ώστε οι αγορές να έχουν μεγάλη αγοραστική δύναμη και να συμβάλλουν στα ταμεία συνοχής. Ε, Σωστός, σωστή στοχοθέτηση και απορρόφηση των ε, ταμείων συνοχής θα βοηθήσει την Ένωση να φτάσει στα κατάλληλα επίπεδα ανάπτυξη για σωστή συμμετοχή στην ενιαία αγορά ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του, της Ευρώπης 2020. Οι συστάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμού έχουν στόχο να παγιώσουν να να, να συσπυρώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση με, για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εγώ ακολούθησα την έκθεση του Σελβατόρου Γκαρίγκα, την έκθεση δηλαδή που εγκρίθηκε μέσω του ψηφίσματος 8 Ιουνίου 2011 Όσον αφορά το ΠΔΠ και τους ίδιους πόρους, επίσης έχουμε ψηφίσματα που υιοθετήσαμε τον Ιούνιο φέτος. Στο σχέδιο γνωμοδότησης στην Επιτροπή μας, στις 28 Ιουνίου, εγώ συνέστησα το ποσό των 376 δις για την ε, πολιτική συνοχή, όπως προτείνει η Κομισιόν, ως μήνυμο με επίπεδο χρηματοδότησης για την πολιτική μας, ώστε αυτό να αποτελεί την κόκκινη γραμμή για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις του Κοινοβουλίου για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ θέλω τώρα κάποιες διευκρινήσεις από την Κομισιόν γιατί την περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι έκανε αυτήν την τεχνική ενημέρωση, τεχνική ενημέρωση για το συνολικό ποσό λόγω της Κροατίας, λόγω κάποιων άλλων μακροοικονομικών στοιχείων που ωστόσο δεν είναι σαφής γιατί σύμφωνα με αυτό το έγγραφο ε, λέει ότι για την πολιτική συνοχή θα έχουμε 3 δις 243 εκατομμύρια επιπλέον. Σημαίνει ότι το συνολικό ποσό είναι 379 δις 243 εκατομμύρια. Ε, δηλαδή, Χτες προσπάθησα πραγματικά σκληρά να διαβάσω τη σελίδα αυτή, αλλά δεν κατάφερα να τα καταλάβω ακριβώ τι λέει. Και ε, Επίση, προσπάθησα να έρθω σε επαφή με την Κομισιόν. Πώ είναι δυνατόν, άμα έχει μια τεχνική ενημέρωση λόγω τη διεύρυνση με μια χώρα, την Κροατία, συν κάποια νέα μακροοικονομικά στοιχεία, να έχεις μείον 5 εκατομμύρια στη μια σελίδα και να καταλήγεις ε, τα συν 3 δις για την πολιτική συνοχή. Αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί λοιπόν πριν φτάσουμε στα τελικά στοιχεία. Νομοθετικό πακέτο λοιπόν και είδαμε ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την κοινή μας θέση. Ε, έχουμε ζητήσει μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν ε, την πολιτική συνοχή κατάλληλη στην, ε, για την Ένωση, ε, πιο αποτελεσματική και πιο διαφανή για τους δικαιούχους, ευκολότερη στη διαχείριση από πλευρά των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Αυτό είναι ο στόχο τη επιτροπή μας εδώ. Και οι προτεραιότητε αυτέ δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρί, τη σωστή, να υλοποιηθούν μάλλον χωρίς τη σωστή χρηματοδότηση. Και το λέω για να σα θυμίσω την κόκκινη γραμμή όσον αφορά την πολιτική συνοχή στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται να κατεβούμε κάτω από αυτό το ενημερωμένο ποσόν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διευκρινίσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά σήμερα από πλευρά των ε, εκπροσώπων της Κομισιόν. Προσβλέπω και στην γνώμη των ε, συναδέλφων εισηγητών. Ήρθα σε επαφή με τους ε, σκεώδεις εχθές και περιμένω να ακούσω την άποψή τους. Σας ευχαριστώ. Μια Κρίνησε πριν δώσω το λόγο στο Σκιώδη από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Αυτά τα νούμερα που αναφέρατε από τη τεχνική ενημέρωση που σχετίζεται με την Κροατία και τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία, είμαι σίγουρη ότι η Κομισιόν θα αντιδράσει. Πάντω το θέμα είναι ότι πρόκειται για τη μόνη πολιτική στο πολιετέ ε, πλαίσιο που εξαρτάται από το την ποιότητα και από, τους, ε, από τις ποσότητες και από τις προβλέψεις. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, είναι κάτω το κομμάτι της πολιτικής συνοχής. Λόγω της ε, προσχώρησης της Κροατίας φτάνει πάνω από 8 εκατομμύρια, οπότε, δισεκατομμύρια, συγγνώμη. Οπότε η διαφορά που βλέπετε είναι ότι υπάρχουν περισσότερα χρήματα για να ληφθεί υπόψη η Κροατία, 8 δις και 5 δις λιγότερα λόγω των νέων ε, στοιχείων. Η Κομισιόν ωστόσο ε, επιμένει να μείνει η διευκόλυνση διασυνδέοντας την Ευρώπη μέσα στο Ταμείο Συνοχής, ε, οπότε έχουμε το ίδιο ποσό, αλλά στην ε, πρόταση του Συμβουλίου, όπως μας είπε ο Γιάν η διευκόλυνση διασυνδέοντας την Ευρώπη έχει βγει από το Ταμείο Συνοχής. Οπότε το νούμερο είναι 40 δις λιγότερο, αν το λάβουμε αυτό υπόψη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησή του, το οποίο αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε τη συμβολή τη Επιτροπή μα στην ενδιάμεση έκθεση του πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Αν και κατανοούμε του δημοσιονομικού περιορισμού των κρατών μελών, οφείλουμε να επιμείνουμε ότι ο μακροπρόθεσμο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο για επενδύσεις, την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και φυσικά για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, και εδώ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η πολιτική αυτή είναι η μόνη ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξη και ω τέτοια θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη σε όλε τι περιφέρειε τη Ευρώπη. Η πολιτική συνοχή αποτελεί το κύριο μέρο τη απάντηση στην κρίση καθώ συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αξίζει και δικαιούται παρκής πόρου. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όπως αποφασίστηκε ξεκάθαρα στην έκθεση ΣΟΥΡΕ και στο ψήφισμα που εγκρίναμε στην Ολομέλεια του Ιωνίου και με το οποίο ανανεώσαμε τη διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου, η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι το ελάχιστο για μας για την πολιτική συνοχή Εάν θέλουμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη, καθώ η πολιτική συνοχή αποτελεί μια αναπτυξιακή πολιτική, εάν θέλουμε να, βρούμε αποτελεσματικέ απαντήσει στην κρίση, τότε χρειαζόμαστε του πόρου για να το επιτύχουμε. Για την πολιτική συνοχή, σύμφωνα με την έκθεση τη ΣΟΥΡΕ, το ελάχιστο είναι το τρέχον επίπεδο χρηματοδότηση, δηλαδή τα 366.849 δι ευρώ τα 376 δις ευρώ που πρότεινε η Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020 δεν ανήκουν αποκλειστικά σε αυτή την πολιτική. Μόνο τα 336 δις ευρώ διατίθενται στην πολιτική συνοχής, μια και τα υπόλοιπα 40 δις ανήκουν στο πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη. Από τη μεριά μα δεν υποστηρίζουμε αύξηση του προπολογισμού στην πολιτική συνοχή, αλλά διατηρώντα το τρέχον επίπεδο του προπολογισμού και με μια σύγχρονη, θεματικά στοχευμένη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα πολιτική συνοχή, θα πετύχουμε πολύ περισσότερα. Σε αυτή την κατεύθυνση προτίθεμε να υποβάλω ορισμένε τροπολογίε, οι οποίε πιστεύω θα ενισχύσουν το μήνυμα που θέλει να στείλει η Επιτροπή μα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική συνοχή στο πλαίσιο του περχόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα του υπόλοιπους κοιόδες που δεν βλέπω. Φρανσουά, θε να μιλήσει εσύ, Αλφονσί? Όχι. Ο Λάμπερτ Φανίστεροι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω εγώ την ε, γνωμοδότηση. Την έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε, δεν είναι καινούρια. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε, πού θα καταλήξουμε με αυτή την ιστορία, πού το πάμε, εν πάση περιπτώσει. Ε, το ψήφισμα για το PDP ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρο πέρσι, ε, την, προ... την περασμένη φορά, εν περιπτώσει, με τίποτα μέσα και τίποτα δεν άλλαξε. Και τώρα πού το πάμε ακριβώ, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, Πρόεδρε. Πότε θα έρθει η στιγμή που θα πούμε στην Ολομέλεια, Ιδού, ε, φέραμε μία ενδιάμεση έκθεση ας πούμε. Πότε θα το ψηφίσουμε αυτό το πράγμα διότι τώρα ακούμε ένα τον άλλον και λοιπόν τα έχω χαμένα. Μπορεί κανείς να με βοηθήσει. Χτες κάναμε μια πρόοδο. Με ψηφοφορία ορίσαμε την πρώτη εντολή. Και κάνουμε κάποια πράγματα για να είμαστε αποτελεσματικοί με τα λεφτά που έχουμε ή που θέλουμε, εν πάση για την επόμενη περίοδο. Και πριν από λίγο δημιουργήσαμε νέα μέσα. Δεν επιχορηγούμε απλώς, δεν επιδοτούμε, αλλά δημιουργούμε και ε, αποτελέσματα μόχλευσης. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ε, μια εξυγχρονισμένη πολιτική συνοχής. Λοιπόν, είναι εξυγχρονισμένη, δεν είναι η κλασική μορφή συνοχή, είναι και ολοκληρωμένη, έχει και στόχου, έχει και αναφορά. Το έχουμε εξυγχρονίσει αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Ε, Ποιο το είπε προηγουμένω, ο κύριο Κόβατσεφ. Είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε στην πράξη όλα αυτά. Ποιος μπορεί λοιπόν να μου πει τι θέλουμε τώρα, πότε θα το φέρουμε στην Ολομέλεια, το Σεπτέμβρη. Πρέπει όλες οι επιτροπές να έχουν ετοιμαστεί. Ξέρω μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Για να έχουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και το έγγραφο τον Οκτώβρη στην ψηφοφορία. Πώς πάει αυτό χρονικά. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Θέλει το λόγο για αυτό το θέμα, αυτή τη γνωμοδότηση πολύ σύντομα. Εγώ τι ξέρω. Ε, η ενδιάμεση έκθεση θα ψηφιστεί. Τώρα το ελέγχω στην ατζέντα μου. Νομίζω τον Οκτώβρη. <gasps> Δεν έχει αλλάξει <laughs> για την Ολομέλεια. Τον Οκτώβρη. Τι λες Λάμπερτ. Μα πώς προετοιμαζόμαστε για αυτό το πράγμα. Ενδιάμεση έκθεση γενικώ ε, δεν λειτουργεί. Εμείς προετοιμαζόμαστε, έτοιμοι είμαστε. Τι θα, θα το ξαναφέρουμε πέντε φορές αυτό το θέμα προσυζήτηση. Για ποιο θέμα μιλάς τώρα, αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση στην ενδιάμεση. Εγώ πώς έχω κατανοήσει τώρα τη διαδικασία. Όλες οι ενεχόμενες επιτροπές που γνωμοδοτούν για αυτά τα θέματα του προϋπολογισμού εργάζονται, όπως εδώ ο Αντρέη Κόβατσεφ, και κάνουν γραμματοτήσεις τις οποίες θα καταθέσουν στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού, που θα ψηφίσει μάλλον το Σεπτέμβρη, τουλάχιστον έτσι μαθαίνουμε, και τον Οκτώβριο θα έρθει στην Ολομέλεια. Άρα, η δική μας γνωμοδότηση θα πάει στην ενδιάμεση έκθεση, στο Λαμασούρ, εν πάση περιπτώσει, στην Επιτροπή Προπολογισμών ε, που είναι η διάσκεψη των Προέδρων. Αυτή την ενδιάμεση έκθεση την κάνει η Επιτροπή Προπολογισμού, δεν την κάνουμε εμεί. Ναι, εντάξει, αλλά οι ημερομηνίε είναι ορισμένε. Πότε θα ψηφίσουμε. Α, όχι τώρα. Πρέπει να ψηφίσουμε εμεί το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτή είναι η συνήθι διαδικασία. Έτσι πάνε στην Ολομέλεια αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ε, ε, ε, Στο μεταξύ θα μεσολαβήσει μια μεγάλη διάσκεψη. Νομίζω 31η Αυγούστου ή 30 Αυγούστου μας είπε χτες ο Υπουργός ο κύριος Μαυρογιάννης ότι θα συνεδριάσει το άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και θα προσκληθούν και οι συγητές από το Κοινοβούλιο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Σήμερα. Επίσης η ενδιάμεση έκθεση θα σέβεται τις συνθήκες, το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή για το PDP ε, ε, δεν θα έχει και τα ποσά και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το γενικό κανονισμό, το σχέδιο γενικού κανονισμού που έχει υποβάλει πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα την ενημέρωση. Το σημαντικότερο είναι για το σχέδιο κανονισμού τα ποσά. Συν η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Έτσι και αυτό δεν είναι σημαντικό. Δεν καλύπτει μόνο την πολιτική συνοχή, αλλά ευρύτερα και την ανάπτυξη πέθρου και την αλία. Στι δικέ μας τώρα τροπολογίες, αυτό έχει σημασία, γιατί η δικιά μα νομοδότηση είναι πολύ μετριοπαθής. Ένα αριθμητικό στοιχείο έχει. Αλλά έχετε την ευκαιρία εσείς για ε, δύο μέρες τώρα και πολιτικές ομάδες και προσωπικά να δείτε αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα και να διευρύνετε ε, αυτό το πλαίσιο ε, πέραν του ενός ποσού. Απλώς σκεφτείτε το εξής. Μην κάνετε σχόλια για αυτό που συζητάει διαπραγματευτικά τώρα το Συμβούλιο, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεχόμαστε αυτή την προσέγγιση και θέλουμε να κάνουμε και τροπολογίε και εκινούμε από αυτή την αφετηρία. Όχι, να το αγνοήσουμε στη γνωμοδότησή μα αυτό. Τουλάχιστον αυτό είναι η δική μου πεποίθηση, αλλά μπορεί και να ασφάλω. Η Κρέλ, συγγνώμη, επειδή καθυστέρησα, βγήκα λίγα λεπτά, αλλά έχω μια ερώτηση. Άκουσα διάβασα την γνωμοδότηση μάλλον του κυρίου Κόβατσεφ και εγώ πιστεύω ότι βασίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά εμείς θα πρέπει να βασιστούμε στην έκθεση Γκαρίγκα και όχι στην πρόταση του προϋπολογισμού της Επιτροπής. Εγώ το κατάλαβα λάθος ή εσείς αλλάξατε θέση. Αντρέη, Μα η πρόταση της Επιτροπής είναι η έκθεση Γκαρίγκα. Μάλλον όχι, δεν ξέρω αν είναι το ένα ή το άλλο. Εμείς λέμε ότι έχουμε κόκκινη γραμμή και δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε από τις ε, ε, αναθεωρημένες και ενημερωμένες προτάσεις συνοχής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να υπολείπονται να, να, ε, των όσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η θέση του Κοινοβουλίου και αφετηρία είναι η έκθεση Γκαρίγκα. Το λέω και όλα στη γνωμοδότηση ότι αυτή είναι η δική μας βάση. Θα πρέπει να έχουμε και κόκκινες γραμμές. Να πούμε μέχρι εδώ και πιο κάτω αποκλείεται. Άλλα σχόλια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για τις τροπολογίες, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε και στις πολιτικές ομάδες να δούμε, να το μελετήσουμε αν θα πρέπει να προσθεθεί τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου και με ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι η ενδιάμεση έκθεση θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια. They confirmed it So if no other comment, I would like to ask αν δεν έχουμε άλλο σχόλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια Ευρωπαϊκή απουσιάζει. Καλά. Ή όχι. Θέλετε το λόγο. Ναι, αλλά εσείς είστε της Περιφερειακής Γενικής Διεύθυνσης, όχι του προϋπολογισμού. Ο κύριος Όμπριχτ, ίσως. Είναι στο 1α ή στο 1β το, το CF. Μα τεχνική έχουν κάνει προσαρμογή μόνο στο νέο σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για το PDP, το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, και τα στοιχεία βάσει της νέας πρόβλεψης, οπότε, που είναι η Κροατία, και κάτι για την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, γράφει εκεί. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Όχι. Yeah, για την ε, ε, επανένωση της Κύπρου. Κάτι γίνεται μνήμα εκεί. Το σημαντικότερο όμως είναι οι αλλαγέ που έχουν γίνει. Η Κροατία είναι η ουδέτερη δημοσιονομικά. Υπάρχει ε, μια πρόβλεψη για phasing in, για σταδιακή ένταξη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει αυτό να το σχολιάσουμε. Αυτό που έχει για μας σημασία είναι τα γενικά ποσά. Α, τώρα όμως είναι έτοιμη να πει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας εκφράζω την λύπη μας γιατί δεν μπορέσαμε να έρθουμε όταν έπρεπε αλλά γραπτός και αποσιοποιητικά. Δεν έχει σχόλια λοιπόν η Κομισιόν, ο Γιάννη Όλμπερτ. Μα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας δοθεί γραπτή απάντηση, αλλά ας θέσουμε το ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. αποσαφήνιση και δεύτερον τα 40 δισεκατομμύρια θα μπουν στην, πολιτική συνοχή ή όχι. Γραπτός καλύτερα. Ναι, γραπτός. Γιατί στην τεχνική ενημέρωση του σχεδίου κανονισμού η Κομισιόν δεν άλλαξε τη δομή, την κατανομή τεχνική προσαρμογή έκανε το CEF όπως και πέρυσι είναι μέσα στην πολιτική συνοχή. Ναι, αυτό είναι στα έγγραφα της Κομισιόν, αλλά ε, ξέρουμε από άλλες πηγές ότι υπάρχει και το Συμβούλιο που μπορεί να διαφέρει. Άρα γραπτός να μας πει η Κομισιόν τι συμβαίνει σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν σχέδια αλλαγών. Ε, με αποσαφήνει σούλα. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε επισήμως από την Κομισιόν Ελπίζω να μην χρειάζεται επιστολή εκ μέρους μας, αλλά να αρκεί να μας πείτε ότι θα μας δώσει γραπτή αποσαφήνιση η Κομισιόν ως προς το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Νομίζω ότι θα απαντήσετε ότι δεν αλλάζει τίποτα, αλλά να το έχουμε γραπτό να το μεταβιβάσετε αυτό το αίτημά μας στην Κομισιόν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια για το ίδιο θέμα. Μήπως Ανδρέα θέλεις να αντιδράσεις. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα περιμένω τις τροπολογίες τις επόμενες ημέρες. Α Ίσως την επόμενη εβδομάδα και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους Κιώδης για να καταλήξουμε σε ένα σωστό και στεναρό κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Η διορία κατάθεσης τροπολογιών θα λήξει το πολύ στις 17 Ιουλίου το μεσημέρι. Την Τρίτη δηλαδή. Ευχαριστούμε. Πάμε πάλι στον Μάρκους αφού ήρθε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή του. Δεν ξέρω αν ήρθε ο Βίκτορ Μποστινάρο. Μόνο ο Σόλτς είναι εδώ από τους κοιόδης. Α, σου είχα δώσει το λόγο, Όλτζι, δεν το κατάλαβες. Ευχαριστώ πολύ για αυτό, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συζήτηση αυτή είναι τρομακτικά ε, σημαντική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλες τις πτυχές του θέματος και να καταλάβουμε ότι η κατανομή των κονδυλίων είναι αυτή τη στιγμή τρεις φορές υψηλότερη από ό,τι την προηγούμενη περίοδο. Ήταν 12 δισεκατομμύρια και για τα θέματα μεταφορών και ενεργείας Ενώ αν δούμε τώρα την κατανομή για αυτή την περίοδο, τα 10 δισεκατομμύρια περίπου θα χορηγηθούν στο ICT και η τροπολογία μου προβλέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλαμβάνει και τα λεγόμενα έξυπνα δίκτυα για τα ενεργειακά δίκτυα νομίζω ότι η σύνδεση είναι σαφής. Είναι δύσκολο να προφηθούν τα κονδύλια αυτά λόγω όλων των αδειοδοτήσεων που χρειάζονται τις άδειες δημιουργίας δικτύων κλπ όλους τους όρους που προβλέπονται καθιστούν πολύ δύσκολη την πραγματική χρήση κατά την ψηφοφορία εγκρίναμε μία τροπολογία που αφορούσε τη μεταφορά 10 δισεκατομμυρίων από την πολιτική συνοχής και καταλήξαμε στο συμβιβασμό που έλεγε ότι για ολόκληρη την επόμενη προγραμματική περίοδο τα χρήματα από την πολιτική συνοχής για το CEF θα συνεχίσουν να είναι τμήμα της εθνικής κατανομής ή θα συζητιούνται διμερώς μεταξύ του κράτους και της Κομισιόν. Αυτό νομίζω πρέπει να το κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση, ώστε να είναι όλα σαφή και να ξέρουν όλοι τι συμβαίνει. Επίσης πιστεύω ότι για να είμαστε πιο ευέλικτοι και ευέλικτες Πρέπει τα προγράμματα αυτά να διευρυνθούν ως προς τουλάχιστον το τμήμα που αφορά τις μεταφορές με διαπραγματεύσεις από τα κράτη-μέλη με καλύτερη ευελιξία και να δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη περιφερειακές ή τοπικές πραγματικότητες. Το επόμενο τεχνικό μου σχόλιο αφορά την ενέργεια, το τμήμα που αφορά την ενέργεια όπου θα ήθελα να υπάρξει μια αλλαγή από τα λεγόμενα μέτρα χαμηλού διοξιδίου σε μέτρα χαμηλών εκπομπών. Αυτά ζητάει η ομάδα μου. Ο Βίκτορ Μποστινάρου. Ευχαριστώ, συγγνώμη που καθυστέρησα την προσέλευσή μου. And quote uh, from Mr. Uh, Θα αρχίσω από την αρχή. Εχθές ίσως τα μπερδέψαμε γιατί Cohesion Fund Regulation we have adopted a compromise which stipulates είπαμε κάτι που κατέμε για το Connecting Europe τουλάχιστον πρέπει να πούμε τα πράγματα σαφέστερα, να ξέρουμε ποια είναι η βάση, η κύρια αρχή για την εφαρμογή του Connecting Europe. Μπορεί να μην είναι πρόκειτο για λάθος αλλά για συμβιβασμό, αλλά δεν μπορεί η Επιτροπή μας στο σύνολό της να εξαμαρτήσει δις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ για το σχόλιο του. Τα εξακρίβωσα όλα αυτά και αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πιο αμφιλεγόμενο θέμα ανέκαθεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθούν τα 10 δισεκατομμύρια ή δεν θα μεταφερθούν στην κεντρική διαχειριστική αρχή. Άλλο σημαντικό θέμα που λύθηκε από τον χθεσινό συμβιβασμό αφορά τον λόγο που έχουν τα κράτη της συνοχής για τα προγράμματα που πρέπει να εφαρμοστούν σε σχέση με το Connecting Europe. Και σας ξαναλέω ότι ο χθεσινός συμβιβασμός είναι σημαντικός και είναι θετικός και για το Συμβούλιο και για την Κομισιόν. Ο χθεσινός συμβιβασμός προέβλεπε να μην μεταφερθούν τα χρήματα, να κρατηθούν στο, στην εθνική κατανομή και πριν από κάθε εφαρμογή η κεντρική διαχειριστική αρχή να έχει πρώτα να πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους. Αυτό νομίζω είναι θετικό και σωστό γιατί επιτρέπει την εφαρμογή του προγράμματος αλλά με τις απαραίτητες εγγυήσεις. Φυσικά υπάρχει ακόμη εδώ χώρος για διαπραγμάτευση, περιθώριο. Αλλά το ίδιο πρέπει να ισχύει και αλλού. Και για το Connecting Europe ιδίως. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό για μένα η ιδέα της πρόβλεψης του 30% του Connecting Europe για σχέδια διαμεθοριακού χαρακτήρα. Καταρχάς, το Connecting Europe έχει όντως μια τέτοια διάσταση και είτε πρόκειται για την ενεργειακή πτυχή είτε για τις υποδομές των μεταφορών αλλά Ίσως 30% να είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Και οι λόγοι του καθορισμού του δεν έχουν εξηγηθεί πλήρως από τον εισηγητή. Πρέπει να βάλουμε μεν κάποιο ποσοστό τμήμα για το σκοπό αυτόν, αλλά όχι 30%. Γιατί είναι πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα αλλά και άλλες που έχουν λιγότερο κρίσιμα προβλήματα. Το ποσοστό λοιπόν αυτό μειώνει δραστικά την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται. Βρισκόμαστε σε πρώιμη ακόμη φάση. Μετά από το σχέδιο έκθεσης θα δούμε τις τραπολογίες αλλά θα ήθελα να δηλώσω προς τον εισηγητή και όλους τους υπόλοιπους που ενδιαφερόμενους, Συμβούλιο και Επιτροπή, ότι τέτοια προγράμματα προφανώς είναι σημαντικά. Όντως χρειάζεται το Connecting Europe, αλλά επειδή υπάρχει και αντίθεση, ξέρετε κυρία Πρόεδρε ότι υπήρχαν 20 τροπολογίες πλήρους διαγραφής του Connecting Europe. Υπάρχουν διαμάχες και μέσα στο Συμβούλιο. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει συμφωνία για να εφαρμοστεί το Connecting Europe, τότε θα έπρεπε όλοι μα όλοι να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτά τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για να επιτευχθεί γιατί αν αυξηθεί η αντίθεση τότε μάλλον θα κινδυνέψει και η ίδια η ύπαρξη του Connecting Europe. Πρέπει λοιπόν να συνδυαστούν, να συμφιλειωθούν οι δύο απόψεις και ελπίζω το φθινόπωρο μετά τας διακοπάς και η DG Move η Move θα καθώς και η Επιτροπή Μετάφη δική μας θα λάβει υπόψη της την ανάγκη να υπάρξει συμβιβασμός. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, ελπίζω και οι άλλοι να το πράξουν, διότι τελικά θα ισχύσει ό,τι από κοινού συμφωνήσουμε. Πρέπει να καταλήξουμε στο συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Ο Λαμπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ Μάρκος. Εδώ έχουμε την ε, το θέμα, μια παροιμία λέει ότι στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Εχθές τι αποφασίσαμε. Σαφές. Υποστηρίζουμε τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη ισχυρά, στεναρά, ε, γιατί τα μέσα που είχαμε στο παρελθόν δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά για να ρυθμίσουμε αυτά τα δε συνοριακά ζητήματα. Και εμείς και το θέμα της ανάπτυξης και αυτά όλα περί της ε, ενέργειας και των στόχων. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε θα πρέπει να είμαστε πιο εστιασμένοι και γεωγραφικά ευρύτερα χρειάζεται οπωσδήποτε μια προσαρμογή και προσέγγιση. Εχθές όμως είπαμε ας το κάνουμε αυτό βήμα-βήμα. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει πραγματική διευκρίνηση, και δεν είναι και τόσο δύσκολο πιστεύω, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε ερωτήσεις που έκανε ο Γιάνν Όλμπριχτ και ο Μάρκους στα πλαίσια του PDP. Για πούμε, για έλα εδώ λοιπόν κυρία Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας τα λύσεις αυτά. Πού θα μπουν, στη συνοχή ή εκτός συνοχής. Και τι και αυτό λογικό είναι. Κάνετε μια πρόταση για μια λύση, όχι. Τούτη τη βδομάδα πήραμε ένα κείμενο σούπα. Ό,τι θέλετε είχε μέσα και γεμάτο ασάφειες. Γι' αυτό ψηφίσαμε χτες για να έχουμε μια πάρα πολύ σαφή προσέγγιση και παραμένουμε πραγματικά στη γραμμή της συνοχής. Και αν δεν το αυξήσουν αυτό, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από εκεί τα χρήματα. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Μποστινάρου και στη δική του έκθεση, εμείς είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε, αλλά δεν κάνουν βήματα προς την πλευρά μας. Αν θέλουν να μας πείσουν, ας έρθουν δύο επίτροποι παρακαλώ εδώ στην Επιτροπή να μας τα πούν. Είμαστε συνομοθέτες. Για ελάτε παρακαλώ να μας πείσετε αν θέλετε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν το προσάπτω αυτό στο Μάρκος. Λέει ο Μάρκος, εντάξει, μπορεί να ε, υιοθετήσουμε ένα από τα άρθρα που δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ε, ε παραπέρα ο Μάρκος σε σχέση με αυτά που εμείς χτες αποφασίσαμε στην ψηφοφορία. Αλλά να δούμε. Εγώ δεν βλέπω ακριβώς την ε, αντίφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα διευκρινίσει αυτά. Ας πούμε στην παράγραφο 15 λες ε, ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα του κάπινγκ, δηλαδή της οροφής. Ε, να μας τα εξηγήσει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά, να καταλάβουμε τι θέλουν. Το μπαλάκι είναι στη δική τους πλευρά και χτες στην ψηφοφορία μας ε, και μετά την ψηφοφορία αρχίσαν τα τηλεφωνήματα. Γιατί τα ψηφίσατε αυτά. Δεν διαβάσατε τι ψηφίζετε. Δεν διαβάσατε το έγγραφο εργασίας. Είπαμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε και η Κωνσταντσα και να βάλουμε και περισσότερους μοχλούς από τις άλλες φορές. Και θυμηθείτε παρακαλώ, πέρσι το Νοέμβρη καταθέσαμε το έγγραφο εργασίας και έκτοτε ψυγεί ηχθείως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς έχουμε τις ευθύνες μας, τις αναλαμβάνουμε, Πώ το λένε αυτό για τη συνδιαχείριση και τα λοιπά. Λοιπόν, διευκρινίζω ότι χτε δεν ψηφίσαμε λάθο στην ψηφοφορία, όχι, λάβαμε θέση. Ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση, διότι η εντολή είναι διαπραγματευτική. Και αν γυρίσουμε και σα πούμε ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση και πανευτυχή, ωραία. Όπω προτείνει λοιπόν ο Μάρκο, θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά θέλω να κινηθεί και άλλη πλευρά της ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερος. Συμφωνώ πολύ με τον Μάρκος να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στις ε, διασυνοριακές συνεργασίες και με ποσοστά συγκεκριμένα, μάλιστα και χτες συγκεκριμένα αποφασίσαμε. Ε, και ένα τελευταίο. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Νότια Ευρώπη με όλα τα δεινά και με τη διασύνδεση και με όλη την ηλιακή ενέργεια που αν θέλουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στη Βόρεια Ευρώπη. Και πού είναι η νέα οικονομική δραστηριότητα και η αναζωγόνηση της οικονομίας τους. Το υποστηρίζω λοιπόν αυτό. Και ένα τελευταίο, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έρθει με συγκεκριμένη πρόταση για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, θα καταπέσει το σύνολο θα γκρεμιστεί. Δεν είναι ότι ζητάω εγώ διευκρινήσεις. Οι ίδιοι διακινδυνεύουν το όλο εγχείρημα, διότι σε τελική ανάλυση, αν διαβούμε το Ρουβίκονα, δηλαδή το Συμβούλιο, στη συζήτηση του Συμβουλίου θα καταρρεύσει λοιπόν. Έλα λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πού είσαι, βιάσου εν πάση περιπτώσει. Just before I give the floor. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στο Γιάννη, θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάποια παρατηρήσει. Στι 12 Ιουνίου έστειλα τέτοια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούσα διευκρινήσει. Δεν σου απάντησαν. Όχι, όχι, δεν έχει περάσει και πολλή χρόνο, μόνο ένα μήνα έχουμε από τότε. Ε, Γιάννη. Yes, ε, ε, ε, I think that... Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε με την θέση μας ως Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και ακριβώς τι τρέχει. Καταρχήν υπάρχει η πολιτική ανάγκη για να δημιουργήσουμε ένα, ένα μέσο που θα μας επιτρέψει να έχουμε ε, κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενέργεια ε, και τις μεταφορές, ε, πληροφόρηση και αυτά αναφέρθηκαν από την Κομισιόν. Τα 50 δις, 40 συν 10, όχι τυχαία, μπήκαν στο 1β στην πολιτική συνοχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή ότι μπήκαν αυτά τα χρήματα στην πολιτική συνοχή και αυτή εξορισμού βασίζεται στην κοινή ε, διοίκηση, shared management, διαχείριση, συνδιαχείριση. Ε, μέθοδος είναι να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ή να χρησιμοποιήσουμε έναν υπάρχοντα οργανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να βρούμε ε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό είναι ένα είδος δράσης, είναι όπως τα TNT, ε, τα διευρωπαϊκά που, δίκτυα που είναι βασισμένα στις Βρυξέλλες. Εγώ νομίζω Τώρα το αν θα είναι και νέο, νέα, νέος οργανισμός ή όχι είναι ένα ανοιχτό θέμα, αλλά δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Το δεύτερο θέμα είναι, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν θα είναι δυνατόν να μπει αυτό στο έγγραφό μας. Είναι το θέμα των οροφών, του κάπινγκ. Γιατί το κάπινγκ δεν υπάρχει σε κανένα κανονισμό. Αυτό είναι θέμα πολιτικής συμφωνίας από τα κρατημέλη και την Κομισιόν η Κομισιόν πρότεινε το κάπινγκ στο σημείο 5 είναι υποσυζήτηση διαρκώ στο PVP στο 2,5% με συγχωρείτε και ε, θέλει να βάλει ε, την οροφή σε ολόκληρο το Ταμείο Συνοχής. Μας αρέσει, μας αρέσει, το κάνανε δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο κείμενο ενός ε, ε, νομικού κανονισμού εφόσον πρόκειται μόνο για πολιτική συμφωνία. Δεν πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για κάπινγκ γιατί δεν είναι θέμα ε, νομικό, είναι η συζήτηση για το PDP. Και το επόμενο στοιχείο είναι το Ταμείο Συνοχής βέβαια. Όλοι μας ξέρουμε, εδώ και μήνες, και μήνες το ξέρουμε, ότι μια επιτροπή λέει ότι, ότι τα χρήματα τα, τα παίρνουμε, ενώ ο άλλος επίτροπος λέει ότι τα, τα χρήματα τα δίνουμε. Και το, αυτό το παραθέτω. Είναι τα λόγια των επιτρόπων. Και η έκκληση του Λάμπερτ είναι ξεκάθαρη. Αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό για μας αυτό, αν τα παίρνουν, τα δίνουν είναι το πρόβλημα του συστήματος της πολιτικής συνοχής. Έχουμε ένα σύστημα που λέει ότι το Ταμείο Συνοχής είναι για τα μεγαλύτερα προγράμματα και βασίζεται στα, στη συνθήκη του Μάστριχτ. Αυτά σύμφωνα με τις μακροοικονομικές κυρώσεις και έχουμε το παράδειγμα της Ουγγαρίας. Αν έχουμε λοιπόν το Ταμείο Συνοχής το ίδιο και επανεισάγουμε και έχουμε, έχουν μειωθεί κάποια χρήματα από εκεί και τα χρήματα μεταφέρονται κάπου αλλού, το θέμα είναι θα εξακολουθούν να, είναι ταμείο συνοχή ή όχι. Η απάντηση που πήραμε από την Κομισιόν είναι ότι δεν θα είναι πια χρήματα του Ταμείου συνοχή. άρα θα μειωθεί το Ταμείο συνοχή. Θα είναι είδο χρημάτων του Ταμείου συνοχή με τη σύγχρηματοδότηση που είναι καλό για τον τελικό δικαιούχο, αλλά δεν θα είναι Ταμείο Συνοχής γιατί δεν θα είναι ε, δεν θα έχει μακροοικονομικές κυρώσεις. Δηλαδή, προετοιμάζουμε ένα σύστημα και στη συνέχεια μειώνουμε τα χρήματα. Κατά τη γνώμη μου, κάποιος έχει κάνει λάθος. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν, να είχαν μπει κάποια χρήματα στην άκρη. Τώρα όμως, <clears throat> εγώ είμαι σταθερά κατά του να αφαιρεθούν χρήματα από το Ταμείο Συνοχής γιατί δεν έχει αυτό να κάνει, καμία σχέση με το, προ, με το σχέδιο και τα σχέδια είναι σωστά ή αλλιώς να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα σχέδια αυτά, τα προγράμματα. Έγινε και πρόταση για αλλαγή ενός του προγράμματος. Μπορούμε να αλλάξουμε και τη λίστα των προγραμμάτων. Είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορούμε να συζητήσουμε για το κατά πόσο είναι σωστά όλα τα προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι κατά του να φύγουν αυτά τα χρήματα, τα δέκα δις. Αλλά θα το στήριζα να, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα, αλλά με διαφορετικό τρόπο, όπως με το earmarking, υποχρέωση ή, κάτι, ή κάποιο ομόλογο, ή κάτι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αν τα χρήματα φύγουν, μετά θα αρχίσουμε το, το πληστηριασμό. Όποιο έρθει πρώτο παίρνει τα περισσότερα, ποιο, όποιος είναι καλύτερο πάλι παίρνει τα περισσότερα είναι ασαφές τελείως το μήνυμα. Όποιος προλάβει το κύριο είδε βασικά. Άμα δεν είναι όμως αυτό ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκό σύστημα. Τελευταία μου παρατήρηση. Έχετε παρατηρήσει ότι σε όλα τα, ε, τα έγγραφα που δουλεύουμε τώρα δεν υπάρχουν νούμερα. Είναι το μόνο έγγραφο που συζητάμε με νούμερα. Μα πώς γίνεται. Βάζουμε χ, χ, χ παντού. Ε, πώς μπορούμε να συζητάμε για τα 10 εκατομμύρια και αν έχουμε μείωση του Ταμείου Συνοχής, πάει κάτω δηλαδή, θα είναι ακόμα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή θα είναι παραπάνω από ό,τι πριν. Ας βάλουμε χ, χ, χ, χ, άγνωστος χ. Δεν πειράμε να μιλάμε για 10 εκατομμύρια για το Ταμείο Συνοχής, γιατί αν μειωθεί, καλύτερα να, να μην βάλουμε νούμερα είναι αδύνατο να δουλέψουμε έτσι. Συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά... Λοιπόν, πρώτον, στηρίζω το Ταμείο Συνοχής. Όχι, τη διευκόλυνση. Τη διευκόλυνση, συγγνώμη. Συνδέοντας την Ευρώπη δεν έχω πρόβλημα με τα 40 δις πώς θα κατανοηθούν. Η Κομισιόν θα έχει το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι ένας στόχος. Αλλά νομίζω ότι το να αφαιρεθούν χρήματα από το Ταμείο Συνοχής θα πει ότι καταστρέφουμε το σύστημα. Καταστρέφουμε το σύστημα γιατί ποια θα, τι θα γίνει στην πράξη. Τα χρήματα θα βγουν από το Ταμείο Συνοχής, θα βγουν στην υπηρεσία, στην οργανισμό. Μετά τα κάτι μέλη θα ζητάνε τα λεφτά από τον οργανισμό και μετά θα πρέπει να κάνουν το πρόγραμμα εκείνα να το υλοποιήσουν. Γιατί το πρόγραμμα δεν το υλοποιήσει ο οργανισμός αυτός, θα είναι πάλι τα κρατημέλη, απλά θα προσθεθεί ακόμα ένα βήμα. Εγώ είμαι κατά λοιπόν του να αφαιρεθούν χρήματα από το Ταμείο Συνοχής. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Ζέμπερ. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τα όσα είπε ο Γιάννα Ολμπρίχτ, θα πρέπει να πούμε ότι γενικά ε, στο σύστημα θα πρέπει να ε, λυθούν οι αδυναμίες και χρειάζεται κάποιος κεντρικός συνδυασμός και σχεδιασμός. Ε, πρόκειται για διασυνοριακή συνεργασία με ένα ωραίο δίκτυο ε, είναι σημαντική η διασυνοριακή συνεργασία για την εσωτερική αγορά. Λείπουν και οι επενδύσεις ε, και τα χρήματα και η βούληση. Ας πούμε κάποιος φτιάχνει ένα αυτοκινητόδρομο ή ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, μια γραμμή, σταματάει στα σύνορα και μετά το χάος. Και η πρόταση του Μάρκους Πίπερ ε, προσφέρεται εδώ να κάνουμε μια πρόοδο και ιδιαίτερα χαίρομαι για την τροπολογία του ε, ε, υπαριθμών 9 που μιλάει για την οικολογική διάσταση ε, της κυκλοφορίας και των μεταφορών. Για την τροπολογία 12, τώρα που μιλάς για τα συνοριακά έργα και τους κοινού διαγωνισμούς. Κοίτα, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός. Τεχνικά δεν το καταλαβαίνω πάντα διαμαρτύρονται οι αρχές και απευθύνονται σε μένα. Εκεί ισχύουν ε, πολλές ρυθμίσεις, πολλά ε, δίκαια και το ευρωπαϊκό και το εθνικό. Ε, η ιδέα μπορεί να είναι καλή, αλλά στην πράξη αυτό πώς θα γίνει. Ας πούμε, εγώ θέλω να φτιάξω ένα δρόμο. Είναι τελείως διαφορετικέ οι μέθοδοι, οι διατάξει, η υποβολή προτάσεων. Ένα δίκαιο θα πρέπει να ισχύει, δεν ξέρω, το εθνικό, το ε, ευρωπαϊκό, γιατί πραγματικά επικρατεί τεράστιο χάος. Και θέλω να ρωτήσω τέλος και το Μάρκος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάρκεια των διαδικασιών αδειοδότησης. Σε όλα τα μεγάλα έργα, είτε είναι υποδομές είτε είναι ενέργεια, τραβάει σε μεγάλο μάκρος χρονικά 5, 6, 7, 8 και 10 χρόνια διαδικασία να πάει στην άδεια. Ε, στους σιδηροδρόμους, ε, στους αυτοκινητοδρόμους τραβάει σε πολύ μεγάλο μάκρο αυτό. Ο Επίτροπο Σόιτιγκερ έκανε μια πρόταση για τα ενεργειακά δίκτυα και έλεγε το πολύ τριετία. Πολύ θαραλέα αυτή η πρόταση. Γιατί ξέρουμε μέχρι να γίνει μελέτη αντικτύπου περιβαλλοντικού κλπ. χαιρετίσματα. Εδώ δεν λέει τίποτα σχετικά. Δεν θα είχε νόημα να σκεφτούμε να υπάρχει και μια προθεσμία για να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Γιατί αν το 2014 πάρουμε τα λεφτά και τα πρώτα έργα υλοποιηθούν το 2024, ε, είναι πρόβλημα αυτό. Ε, επειδή είναι και περίπλοκο το θέμα, θα πρέπει τα κράτη-μέλη κάπως να πιεστούν να ε, κάνουν μια πιο ε, συγκεντρωμένη διαδικασία με μια ενιαία θηρίδα και μέσα σε τρία χρόνια να είναι έτοιμο το έργο για την κατασκευή του. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Yes, Constanza Constanza Αυτό που είπε ο κύριος Έμπερ με κάνει να πάρω το λόγο για να ξεκαθαρίσω το εξή. Έχετε δίκιο. Και εμείς όλοι εδώ θέλουμε και ο Λάμπερτ και εγώ το έχω υποστηρίξει αυτή τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αλλά εχτες, αν δεν είχαν βρει ε, συμβιβασμό θα κατέρεε, δεν θα υπήρχε καν η διευκόλυνση αυτή, δεν θα τη συζητούσαμε. Γιατί εμπίπτει στο γενικό κανονισμό και ήταν πολλές οι τροπολογίες που ζητούσαν πλήρη διαγραφή, χωρίς κανένα συμβιβασμό. Τελικά βρήκαμε ένα συμβιβασμό, ελπίζω να μπει και στη γνωμοδότηση του Μάρκους Πίπερ και ελπίζω να αρχίσουμε σιγά σιγά να αλλάζουμε νοοτροπία και ε, τακτική. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε ότι τα κράτη ενδιαφέρονται ε, ένα κεντρικό σχεδιασμό και δεν κοιτούν τι γίνεται πέρα από τα σύνορα ή στα σύνορα. Αλλά με τη χθεσινή απόφαση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο και να μην ε, κάνουμε σαν να μην υπήρχε αυτή η χθεσινή απόφαση της ψηφοφορίας. Και στις επιτροπές του Κοινοβουλίου λίγο να κινηθούμε για να διαμορφώσουμε δημιουργικά αυτή τη δυνατότητα και η Επιτροπή Μεταφορών νομίζω μπορεί να την υιοθετήσει και κάπως να σκεφτεί πώς μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο και να τα συνδυάσουμε. Αλλιώς θα έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Κάποια στιγμή θα φτάσει και στην Ολομέλεια και στο Συμβούλιο η συζήτηση, η διαπραγμάτευση. Ε, θα πρέπει να έχουμε και μέτρο, να είμαστε και πρόθυμοι για πρακτικές λύσεις και εφαρμόσιμες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you. Anybody else? Um, I don't know the Commission. Anybody... Ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πακέ. Δεν, δεν βλέπω με τα γυαλιά μου εκεί ποιος είστε. Ε, καλώς ορίσατε πάντως, όποιος και να είστε. Ε, σας ευχαριστώ. Στέφαν Γόκερ από τη Γενική Διεύθυνση MOVE. Δεν μπορούσε να έρθει ο αρμοδιότερος από μένα και τον αντικαθιστώ. Εμείς δεχόμαστε τα περισσότερα στοιχεία της έκθεσης του κυρίου Πίπερ και στηρίζουμε πλήρως την ιδέα της διενίσχυσης της συνέργειας μεταξύ των ταμείων. Το 60% ήδη στην πράξη των κονδυλίων διατίθενται για διαμεθοριακά προγράμματα, άρα δεν βλέπουμε πρόβλημα. Ακούσαμε σήμερα εδώ πολλά ερωτήματα για τα 10 δισεκατομμύρια. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η μεταφορά ή η λεγόμενη μεταφορά των 10 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Συνοχής για το Connecting Europe πρέπει να το θεωρήσουμε ως ένα δημοσιονομικό τέχνασμα. Τα χρήματα δεν έχουν προταθεί για το Ταμείο Συνοχής από την Κομισιόν αλλά από την αρχή για το Connecting Europe. Είναι ένα τέχνασμα το να τα βάλει κανείς πρώτα στο Ταμείο Συνοχής και μετά στο Connecting Europe για το έτσι ώστε τα 10 δισεκατομμύρια να είναι σίγουρο ότι θα πάνε εκεί και γι' αυτό το Connecting Europe επειδή το διαχειριζόμαστε κεντρικά ο μόνος τρόπος να υπάρξει θετική άνηση μεταχείριση υπέρ του είναι τα χρήματα πρώτα να περάσουν από το Ταμείο Συνοχής και να διατεθούν από εκεί. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, για να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί ο υψηλότερος συγχρηματοδοτικός ρυθμός. Αν δεν γίνει μέσω αυτής της μεταφοράς δεν γίνεται πρέπει να σεβόμαστε την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αν προτείνουμε υψηλότερη συγχρηματοδότηση για ορισμένες περιφέρειες, τότε θα θεωρηθεί ότι δεν κάνουμε ίση μεταχείριση και γι' αυτό η συζήτηση του κατά πόσον πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η κοινή διαχείριση και των 10 δισεκατομμυρίων δεν τίθεται εμείς κάναμε μια σαφή πρόταση που βάζει τα 10 δισεκατομμύρια στο Connecting Europe, στο αποθεματικό του Connecting Europe. Και τα κράτη-μέλη μπορούν να το εξατομικεύσουν δημοσιονομικώς. Αλλά το βέβαιο είναι ότι θα σταλούν στο Connecting Europe. Τώρα για την παρουσίαση του προπολογισμού που κάνουμε. Εμείς προτείναμε ως Κομισιόν το Connecting Europe να παρουσιάζεται σαν τμήμα του υποτίτλου της συνοχής. Καταλαβαίνω ότι το διαπραγματευτικών κοιτίων τα διαχωρίζει, αλλά δεν είναι αυτή η πρόταση της Κομισιόν. Εμείς είπαμε να συμπεριληφθεί στην πολιτική συνοχή ως υπότιτλος. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να υπάρχει η ίδια διαχείριση ή κοινή διαχείριση. Είπαμε ότι υπάρχει απλώς κοινό υπότιτλος. Δεν βλέπουμε καμία αντίφαση μεταξύ των δύο και θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι στις αρχές του 90, στις αρχές του Ταμείου Συνοχής τα διαχειρίζονταν τα προγράμματα κεντρικά στην αρχή η Κομισιόν και μετά έγινε η συνδιαχείριση ή κοινή διαχείριση. Επίσης υπενθυμίζω ότι η συνθήκη για τα διευρωπαϊκά δικτύα λέει συγκεκριμένα ότι το Ταμείο Συνοχής μπορεί να χρηματοδοτήσει τέτοια προγράμματα για μεταφορές και γι' αυτό νομίζουμε ότι συμφωνούμε δεν παραβιάζουμε καθόλου τις συνθήκες χρησιμοποιώντας ένα τμήμα των χρημάτων που περνάνε από το Ταμείο Συνοχής για να περάσουν στο Connecting Europe. Άκουσα κι άλλες εναλλακτικές επιλογές για τη χρήση των χρημάτων όπως την πρόβλεψη για συγκεκριμένους στόχους, ιδιαίτερα για διαμεθοριακά λέει προγράμματα. Αυτό το δοκιμάσαμε, δεν δούλεψε, δεν θα δουλέψει και στο μέλλον. Μπορούμε να επανέλθουμε, αλλά ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Οι διαμεθοριακές υποδομές που χρειάζονται τα κράτη-μέλη δεν θα επιτευχθούν. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά και δύσκολα προγράμματα σιδηροδρόμων, ας πούμε, για να υπάρξουν βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον και ποιος θα ζημιωθεί το δυτικό τμήμα που είναι ήδη, έχει ήδη ανεπτυγμένες υποδομές ή οι χώρες συνοχής που τις χρειάζονται. Χωρίς την ύπαρξη αυτής της πιο σύγχρονης υποδομής θα σημειωθούν οι χώρες αυτές. Οι κανόνες του Ταμείου Συνοχής είναι αυτοί που είναι και δεν θέλουμε τελικά οι χώρες μέλη που τα χρειάζονται περισσότερο αυτά τα χρήματα να μην επωφεληθούν από αυτά. Στον Αντιπρόεδρο Κάλλας θα μεταφέρω την πρόσκλησή σας να έρθει να τα εξηγήσει όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν θα αρνηθεί και αυτά είχα να σας πω. Μάλιστα. Θα ήθελα απλώ να σας πω ότι στην Επιτροπή μας εμείς αποφασίζουμε τι θα συζητήσουμε και τι όχι. Όταν μας λέτε λοιπόν να μην συζητηθεί εδώ, διαφωνούμε. Δεύτερον, είπατε ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με χρήματα συνοχής, αλλά απλώ στέλνονται, μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό όμως δείχνει ότι χρειάζονται εξηγήσει από την Κομισιόν. Και θα τα παγώσουμε όλα μέχρι να τις ακούσουμε αυτές τις εξηγήσει γιατί νομίζουμε ότι δεν ακούσαμε την αλήθεια. Τέλος πάντων, να συνεχίσει η συζήτηση. Κωνσταντσα. Ε, ειλικρινά πρέπει να ομολογήσω ότι αν ζούσα στην Ανατολική Γερμανία δεν θα μου συνέβαινε γιατί θα μου βουλευτείς, αλλά θα έλεγα τι είναι αυτά τα πράγματα που μας κάνουν καθοδήγηση, μας κάνετε, ε, μας δίνετε και μαθήματα. Είμαστε βουλευτές, είμαστε στη συναπόφαση, εμείς νομοθετούμε. Συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να κάνει τις προτάσεις, αλλά την απόφαση την παίρνει σε τελική ανάλυση το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Είστε λίγο εκτός θέματος μου φαίνεται. Αυτά μπορεί να τα πει κανείς άτυπα το βράδυ σε ένα δείπνο, αλλά όχι συνεδρίαση επιτροπής, όπου εχθές αποφασίσαμε πράγματα, τα οποία είναι άκρος λογικά. Και έχει ξεκαθαριστεί το εξή. Ο Γιάνν ε, Μπρίχτ έχει απόλυτο δίκιο να ανησυχεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Και θα τον ρωτήσουμε τον Επίτροπο και να έρθει και με τον κύριο Χάν παρακαλώ, όχι μόνος του και δεν θα είναι η τελευταία συζήτηση για αυτά τα θέματα, αλλά μπορεί και για τη διευκόλυνση, συνδέοντας την Ευρώπη, να σας πω ότι τελικά να αναβαγίσει. Δεν ξέρω αν το επιθυμεί αυτό ή είναι επιθυμητό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι πραγματικά δικαιολογημένη ερώτηση και θεμητή. Θα παρακαλούσα λίγο μεγαλύτερη ευελιξία και στη σκέψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θέλει να μιλήσει κανεί άλλο μέλο τη επιτροπή, ο Βίκτορ Μποστινάρ. Been... Πρόεδρε, μα λένε ότι χωρί αριθμητικά στοιχεία, χωρί ποσά, χωρί ιδέα ε, ε, του συνολικού προπολογισμού για τη συνοχή, ποια είναι η μόνη βεβαιότητα, λιγότερο από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό μας είπανε, ότι έτσι κι αλλιώς τα 10 δις είναι είτε μεταφορά από το Ταμείο Συνοχής, είτε δεν θα υπάρξουν ποτέ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πριν οποιαδήποτε και κατάληξη αυτής, ξέρουμε από τώρα ότι θα χάσουμε 10 δισεκατομμύρια. Ε, ε, αυτό είναι παράδειγμα και για την Επιτροπή μας. Ένα αυτό. Δεύτερον, όπως και εσείς και πολλοί, είχα επανειλημμένα προσπαθήσει να ε, πείσω και τους δύο επιτρόπους, και τη Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ και τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, να έρθουν εδώ να προετοιμάσουμε μια κοινή λύση για τη διευκόλυση συνδέοντας την Ευρώπη. Και μέχρι σήμερα αυτή την ώρα που σας μιλάω δεν είχα καμία αντίδραση. Δεν μπορούν να μας εκβιάζουν, αυτό είναι το θέλετε ή όχι. Η ε, συναπόφαση δεν έχει καμία σχέση με το σας κάνει ή δεν σας κάνει. Είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ε, ουσιαστικότατος και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την Κωνσταντζα και όλους τους αγαπητούς συναδέλφους. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο, στο λόγο ο μα μας, Μάρκος Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γελάω με αυτά που ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ με τις εξελίξεις, γιατί συνήθως εγώ είμαι εκείνος που ε, έχει να φέρει όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο για την έκθεσή μου. Κοιτάξτε, ποια μπορεί να είναι η απειλή. Αν καταλήψουμε αυτά τα 10 δισεκατομμύρια για τον οποιοδήποτε λόγο, έχουμε το εξή παράδοξο. Στις πιο πλούσιες περιφέρειες έχουμε 21 δις για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη και είναι και νομικά δεσμευτικό για να απαντήσω στο Ρίχαρτ Σέμπερ. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα να έχουν ολοκληρώσει αυτά τα έργα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή πίεση που κατά τα άλλα θεωρώ πάρα πολύ θετική. Δηλαδή στη Δυτική Ευρώπη θα, θα γίνουν αυτά και θέλουμε πολύ γρήγορα να συνδεθούν και οι αγορές της ανατολική Ευρώπης. Αλλά αν αποτύχει η συζήτηση δεν πρόκειται να συμβούν αυτά τα έργα εκεί. Προσπαθώ λοιπόν εγώ να, φτιάξω, να χτίσω μια γέφυρα. Ομολογώ και παραδέχομαι ότι... Ε, στο άρθρο 48 ο συμβιβασμός 50 δεν με ικανοποίησε. Εγώ θα έλεγα διαφορετικά ότι αυτά τα χρήματα βεβαίω να συνοηθούμε για το πώς θα δαπανηθούν με τα κράτη-μέλη υπό την προπόθεση και τη διαφύλαξη της διαδικασίας ανταγωνισμού. Η διαδικασία ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Αλλιώ έχουμε τύχε Γιάννη, είχα πάντα, business as usual. Καμία επιπλέον πίεση στα κράτη-μέλη για να είναι αποτελεσματικά και θέλω να σχολιάσω αυτό είπε η Ντανούτα και άλλοι. Εδώ και εβδομάδες περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, εγώ το βλέπω αντίστροφα, ότι είναι για μας μια ευκαιρία να κάνουμε προτάσεις, να αναλάβουμε την πρωτοβουλία εμείς. Έκανα την ε, απόπειρα αυτή. Ε, παραδέχομαι ότι δεν είμαι νομικός, πολιτικός είμαι και αρνούμε, Ρίχαρτ, και σε τέτοια θέματα ε, για διεθνείς διαγωνισμούς, για έργα διασυνοριακά να κάνω πρόταση. Δεν μπορώ να το κάνω. Πολιτική ιδέα είναι αυτό που προτείνω. Μπορώ να μιλήσω με την ησυχία μου, σας παρακαλώ. Ε, η ε, εφαρμογή είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πολιτικοί κάνουν προτάσεις για ιδέες. Εκείνοι καλούνται να τις συγκεκριμενοποιούν. Και αυτό έχει να κάνει και με τη διασυνοριακή συνεργασία και τους διαγωνισμούς που προκυρήσονται. Εγώ προσωπικά δυστυχώ δεν είμαι σε θέση να κάνω μια τέτοια πρόταση. Νομίζω ότι απάντησα στο Ρίχαρτ Τζέμπερ έτσι. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους εκείνους που ανησυχούν και φοβούνται ε, Ε, μήπως καταργήσω τίποτα με την έκθεσή ε, Εγώ είμαι δημοκράτη, σημειώνω τα όσα ψηφίστηκαν εκτές με το συμβιβασμό 50 για το άρθρο 48. Αν περάσει αυτό το θέμα του ανταγωνισμού, θα ήμουν ευτυχής. Εγώ τι θέλω, μια διαδικασία σταδιακή. Δηλαδή, ε, όχι ένα διαγωνισμό, ε, προκηρύξεις διαδοχικές και στο μέσο της περίοδου να το ελέγξουμε. Το έχουν ανταποκριθεί τα κράτη στις υποχρεώσεις και να βελτιώσουμε την κατάσταση έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν κάποιοι σε μελλοντικέ προκηρύξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να ασχοληθεί περισσότερο. Εγώ δεν προτείνω και δεν θέλω καθόλου ε, να μείνει πίσω καμία χώρα μέλος και πιστεύω ότι είναι από τα λίγα ε, μέσα στην Ευρώπη που χρειαζόμαστε κεντρική διαχείριση των χρημάτων. Γνωρίζετε ότι εγώ επικρίνω ε, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μάλιστα σφοδρά, αλλά εδώ υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και χρειαζόμαστε κάποια κεντρική διαχείριση. Θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που να μην αφήνει τη συνοχή να χαθεί και να συμμετέχουν και όλες οι χώρες. Τώρα για το κάπινγκ, αυτό την οροφή δεν το καταλαβαίνω. Ε, τυπικά αυτό δεν ανήκει εδώ, αλλά εμείς είμαστε πολιτικοί. Δεν είμαστε ε, ε, τυπολάτρες, πώς να το πω. Μπορεί να μην είναι εδώ η σωστή θέση ε, για τα χρήματα συνοχής ε, με τη διευκόλυνση για την Ευρώπη, αλλά εγώ δεν ήθελα να προτείνω να επιβάλλω τίποτα παραπάνω για τα εκτελεστικά. Τα ξέρει καλύτερα η εκτελεστική επιτροπή αυτά. Και τούτο εδώ το κείμενο είναι γνωμοδότηση απλή μιας επιτροπής. Δεν μπορεί να είναι το απάβγασμα τη Σοφία και τη τελειότητας. Προσπαθώ να βάλω ε, λίγο δυναμικό χαρακτήρα σε μια δύσκολη συζήτηση. Ευχαριστώ Μάρκο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τα χρονοδιαγράμματα τώρα για την έκθεση αυτή, τη γνωμοδότηση μάλλον. Στην Επιτροπή Μεταφορών θα ψηφίσουν 5 Νοεμβρίου. Εμείς μπορούμε τον Οκτώβριο να εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση. Στις 10 Οκτωβρίου, αν δεν απατώμεν, συνεδριάζει η Επιτροπή μας και ε, προηγουμένως συνεδριάζουμε και στις 18 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, αντί να ορίσουμε σήμερα την ε, ε, προθεσμία τροπολογιών. Μπορούμε στις 18 Σεπτεμβρίου να το συζητήσουμε. Ε, γιατί τι να ψηφίσουμε αφού δεν ξέρουμε τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αντιφατικές οι προφορίες που παίρνουμε. Προτείνω στις 18 Σεπτεμβρίου να καλέσουμε την Επιτροπή να δούμε ποιος θα έρθει για να ξεκαθαριστούν τα θέματα και να ορίσουμε τότε τροπολογία. Συγγνώμη, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Αρχίστε από τώρα να το σκέφτεστε για να μην γκρινιάξετε μετά ότι δεν έχουμε χρόνο για τις τροπολογίες και στις 5 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Μεταφορών. Για να κάνουμε καλή ε, γνωμοδότηση χωρίς λάθη. Αν συμφωνείτε. Και τρεις μπορούμε να καλέσουμε, όχι μόνο δύο, όσους θέλετε. Θα δούμε. Θα δούμε ποιο θα Το θέμα είναι ποιο θα καλέσουμε. Ποιοι θα έρθουν στι 18 Σεπτεμβρίου. Αυτά. Τελειώνει αυτό το θέμα εδώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρκους για την παρουσίαση αυτή. Έχουμε άλλε δύο εκθέσει. αγαπητοί συνάδελφοι. Ραμόνα Μανέσκου, η οποία αποσιάζει και δεν έχει ορίσει και κανένα να μιλήσει εξ ονόματός της. Ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Να σας πω λίγο για τις τροπολογίες. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Παπουσία της κυρίας Μανέσκου, τι να κάνουμε. είναι και οι δύο δικές της. Κυρία Ρούλε, ναι, αφού θα αναβληθεί ε, στην ΙΜΚΟ η ψηφοφορία, έχει αλλάξει η μερίσια διάταξη και θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου, 17 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Εσωτερικής. Είσαι, είσαι σίγουρη για αυτά που λες. Ναι, ναι, ναι. Χτες το έστειλαν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ε, της ΣΥΜΚΟ από τη Γραμματεία γιατί το είχαν ζητήσει και ο κύριος Ταραμπέλα και η Σκιώδης. Γιατί πήρε πάρα πολλές τροπολογίες και ζήτησε να αναβληθεί. Άρα μπορούμε να το αναβάλουμε για το Σεπτέμβριο αυτό. Τότε θα φταίσει εσύ αν πάει κάτι στραβά, έτσι, το παίρνει πάνω σου. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τις δύο εκθέσεις κυρίας Μανέσκου για τις δημόσιες συμβάσεις. Θα τις αφήσουμε το έχουμε συνοηθεί με την ΙΜΚΟ. Δεν θέλανε αυτή η αναβολή, αλλά τώρα το αναβάλανε. Τι να κάνουν. Λοιπόν, τότε ερχόμαστε στο τελευταίο θέμα που είναι τα διάφορα. Έχετε κανένα διάφορο, όχι, ε, ούτε εγώ. Ωραία. Προσεχή συνεδρία στις 17 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι και στις 18 και πάλι. Σας ευχαριστώ ειδικά για τη χθεσινή ημέρα. Καλή σας ξεκούραση κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Λήξη συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς. Καλές διακοπές. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ.